So, good morning everybody. Καλημέρα σας. Αρχίζουμε την τελευταία μας συνεδρίαση του 2013. Έγκριση των πρακτικών της ε, προηγούμενης συνεδρίασης. Δεν βλέπω να είναι κανείς ε, αντίθετος. Ε, ελπίζω να συμφωνούμε με την μέρη σε διάταξη δεν έχουμε κάποιες καμπίνες για τη διερμηνία, αλλά επειδή κάποιοι συνάδελφοι λείπουν. Να περάσουμε τώρα στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε το θέμα πολιτιστικές πρωτεύουσες. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε σε πρώτη ανάγνωση την πρότασή μας. Είναι το μόνο σημείο που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε με την ε, Λιθουανική Προεδρία, όχι τόσο πολύ λόγω της Λιθουανικής Προεδρίας, αλλά διότι υπήρχε μια τέτοια συμπεριφορά στο Κορεπέρ που δεν το επέτρεψε. Στο Κορεπέρ θεωρούν ότι ο καθορισμός των πολιτιστικών πρωτευουσών είναι θέμα του Συμβουλίου. Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα ήταν ως εξής είχαμε μία επιτροπή επιλογής εμπειρογνωμόνων που συναποφασίζουμε ε, τα τρία θεσμικά όργανα και με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη κάνει πρόταση η Κομισιόν μέχρι στιγμής την επιτροπή αυτή, την ε, πρόταση αυτή την έστελνε και σε εμά και στο Κορεπέρ δίναμε τη γνώμη μας, μπορούσαμε μόνο να πούμε ναι γιατί δεν ήμασταν εμπειρογνώμονες. Όλο αυτό βέβαια καθυστερούσε γιατί ήταν διαδικασία συναπόφασης και το ίδιο για το Συμβούλιο. Και περνούσε μήνες. Ενώ εμείς μόνο ναι μπορούσαμε να πούμε. Τώρα με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, άλλαξε η διαδικασία. Η Κομισιόν κάνει πρόταση η Επιτροπή Επιλογής καθορίζει τον υποψήφιο, ε, στέλνει την πρότασή της στην υποψήφια πόλη, στέλνει την πρότασή της ε, ε, στην Επιτροπή η οποία την εγκρίνει. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί βεβαίως με αυτή τη διαδικασία και είπαμε ότι εμείς είπαμε ότι αποδεχόμεθα αυτή την στην ουσία διοικητική διαδικασία γιατί κανένα από τα τρία θεσμικά όργανα δεν είναι εμπειρογνώμων. Απλώς αποδεχόμεθα την πρόταση των εμπειρογνωμόνων. Θα θυμάστε, κατά τις διαπραγματεύσεις, δεχθήκαμε ότι το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει συμπληρωματικά δύο εθνικούς εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, δώσαμε σε αυτήν την ε, Επιτροπή Επιλογής ε, περισσότερες αρμοδιότητες. Αλλά δεν το δέχεται το Συμβούλιο, χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Και πέρασαν τόσες εβδομάδες μέχρι να μας κάνει μία πρόταση, την οποία έλαβα Παρασκευή βράδυ. Μου είχαν πει ότι θα λάμβανα αυτή την συμβαστική πρόταση που ήταν πολύ καλύτερη και δεν θα έπρεπε να ε, να ε, αποδεχτούμε να μην υπάρξει πρώτη ανάγνωση. Αλλά εγώ δεν δέχθηκα γουρούνι στο σακί. Κάναμε την πρώτη ανάγνωση. Βεβαίως και η Λιφανική Προεδρία ήθελε να λήξει η διαδικασία, αλλά θα συζητηθεί μόνο αύριο στο Κορεπέρα και είπα ότι εμείς θα δούμε εάν και κατά πόσο ε, συμφωνούμε. Δεν μπορούσα απλώς να το αφήσω αυτό ε, μόνο ε, στο κορεπέρ. Θα ήθελα να ακούσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Και είπα λοιπόν ότι αν κάνουμε αυτή τη ε, διαδικασία θα μπορούσε να αποφασιστεί αύριο. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αύριο στην, ή μεθαύριο στην σε διάταξη του Κορεπέρ και δεν υπάρχει κανείς εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να διοργανώσουμε τριμερή διάλογο με τον ε, συνάδελφο Σίγητη και τους άλλους, γιατί δεν θα είναι πια κανείς εδώ, γιατί είμαστε πολύ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ε, δαπανίσαμε, σπαταλήσαμε 9 εβδομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την Ελληνική Προεδρία τον Ιανουάριο και αν κάποιοι σας πούν ότι το γεγονός ότι θέλουμε να κάνουμε πρώτη ανάγνωση και καθυστερούμε θα οδηγήσει στο ότι οι δύο χώρες που έχουν ε, καταθέσει υποψηφιότητες για το 2020 δεν θα έχουν αρκετό χρόνο. Όχι. Εμείς είπαμε ότι θα έχουν ε, λιγότερη, επιτρέψαμε να υπάρχει ε, μικρότερη προθεσμία για αυτές τις δύο χώρες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα πάνε καλά. Θα τα αναλάβει η Ελληνική Προεδρία πολύ νωρίς τον Ιανουάριο. Ίσως κατά την πρώτη συνεδρία, όταν θα έχουμε τον Υπουργό Πολιτισμού της ε, Ελλάδας, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε μαζί του και με τον εισηγητή για να λύσουμε το θέμα. Ήθελα μόνο να σε ενημερώσει αυτό το θέμα. Είμαι σε επαχή με τον Μάρκος Κορέα και επίσης ε, μας τηλεφωνούσαν για να μας ρωτήσουν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ τους είπα όχι, όλοι έχουμε τις διαδικασίες μας. Εμείς έχουμε μία επιτροπή εσείς έχετε το κορεπέρα. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της μελέτης για το θέμα πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ε, στρατηγικές επιτυχίες και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Έχουμε καλέσει την δόκτωρα Μπεατρίθ Γκαρσία, είναι από το Ινστιτούτο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Θα της δώσουμε το λόγο. Θα ήθελα να μάθουμε εάν είναι σημαντικά αυτά που επιτύχαμε από το Συμβούλιο. Υπενθυμίζω πριν πάρετε το λόγο, καταφέραμε να αποσπάσουμε από το Συμβούλιο στο κείμενο να λέει ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσε θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν ήθελαν να αναφέρεται αυτό. Δεν ήθελαν να υπάρχει και η λέξη ανάπτυξη των πόλεων, αστική ανάπτυξη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι θέματα που τα τελευταία 20 χρόνια τα έχουμε προωθήσει και ήθελα να διαγραφούν όλα αυτά. Γι' αυτό με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω αυτά που ε, θα μας πει η δόκτωρ Γκαρσία. Ελπίζω να μας υποστηρίξει με την εμπειρογνωμοσύνη της και με παραδείγματα. Ε, παρακαλώ κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα η σημερινή μου παρουσία όπου θα σας δω, κάνω την παρουσίαση της μελέτης αυτής της οποίας ηγήθηκα επί ένα χρόνο. Το θέμα βέβαια είναι πολύπλοκο και τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είναι μια έννοια που έχει αποκτήσει αυξημένη ορατότητα η πολιτιστική πρωτεύουσα. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με, σε μελέτες για αυτό το θέμα τα τελευταία 15 χρόνια και ήταν πολύ θετικό ότι μπόρεσα να εξετάσω όχι μόνο περιπτώσεις προηγουμένων πολιτιστικών πρωτεύουσων όπως της Γλασκόβης και του Λίβερπουλ αλλά την όλη εξέλιξη της ενίας. Για πρώτη φορά γινόταν αυτό και ε, καιρός ήταν να γίνει μια τέτοια μελέτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του 12 μας έδωσε την εντολή της μελέτης αυτής για να εξετάσουμε όλα το δημοσιευμένο υλικό για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Πρέπει να σας τονίσω ότι δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε πόροι για μεγαλύτερο, περισσότερο ευρύ ευρύτερη εξέταση των 58 πόλεων που από το 95 μέχρι τώρα είχαν αυτόν τον τίτλο. Θελήσαμε πάντως να συγκρίνουμε ό,τι στοιχεία είχαμε και να ταυτίσουμε τις πιο κοινέ στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει οι πόλεις για να πετύχουν τους στόχους τους. Μαζέψαμε στοιχεία από πολλούς τομείς, όχι μόνο πολιτισμό αλλά και οικονομία κλπ. Για να δούμε ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και προβλήματα. Τώρα ξέρετε, ότι είδατε ότι έχει δημοσιευτεί η μελέτη, έχει μεταφραστεί και η σύνοψή της σε πολλές γλώσσες και θα σας αναφέρω τα κύρια ερωτήματα που θέσαμε στον εαυτό μας και τα μεταφράσαμε σε κεφάλαια της μελέτης από την ιστορία του προγράμματος μέχρι του πώς γίνονταν οι προσφορές που ακολούθησαν μια διαδικασία όλο και πιο επαγγελματική. Θέλησαμε επίσης να δούμε εάν οι στόχοι επιτεύχθηκαν και ποιες ήταν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των εκδηλώσεων. Γιατί δεν είχε νόημα να δούμε μόνον τα αποτελέσματα αλλά να τα συγκρίνουμε και με τις αρχικές προθέσεις για να δούμε αν η διακολουθηθήσα διαδικασία ήταν επιτυχής ή όχι. Γι' αυτό η μελέτη μας καλύπτει όλες αυτές τις πτυχές. Συζητούμε και τα προβλήματα <coughs> και τις προκλήσεις και κάνουμε και μερικές τελικές συστάσεις. Να δούμε το ιστορικό τώρα από την πρώτη εμφάνιση της έννοιας αυτής το 85 μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το τέλος του 19 υπάρχουν τρεις φάσεις. Για να σας τα για να δείτε πόσο πολύπλοκη διαδικασία ακολουθήθηκε από τότε μέχρι τώρα. Οι τρεις φάσεις αυτές λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη ο πρώτος πλήρης κύκλος δηλαδή δώδεκα χωρών μελών εδώ από 12 χώρες μέλη θεωρούνταν η πολιτιστική πρωτεύουσα σαν διακυβερνητική δραστηριότητα χωρίς να διαθέτει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο νομοθετημένο. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο να υποβάλουν οι πόλεις συγκεκριμένες εκδηλώσεις είχαν πολύ λίγο χρόνο για να το πράξουν. Αλλά στη δεύτερη φάση, 97 με 4, για πρώτη φορά διατυπώθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και μπορούσαν οι υποψήφιες πόλεις να περιγράψουν πληρέστερα αυτά που ήθελαν να πραγματοποιήσουν ως στόχους. Και η τρίτη φάση που άρχισε από το 2005 Εκεί είδαμε την εμφάνιση του πρώτου επίσημου νομοθετικού πλαισίου με επίσημα κριτήρια σαφέστερα για τις πόλεις και πιο αυστηρή διαδικασία επιλογής. Σημαντικότερες αλλαγές στην περίοδο αυτή ήταν ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν διευρυνθεί. Πέρα από απλές εορταστικές εκδηλώσεις των πολιτιστικών προσόντων μιας πόλης υπήρξαν και ευκαιρίες να εφαρμοστούν στόχοι και πιο ευρύτερα οικονομικοί. Και οι πόλεις οι ίδιες που έχουν επιλεγεί δεν ήταν μόνον ήδη υπάρχουσες γνωστές πόλεις αλλά και αναδιόμενες πόλεις. Ε, εφόσον διευρύνεται και η Ευρώπη, διευρύνεται και η έννοια αυτή της πολιτιστικής πρωτεύουσας με τη συμπερίληψη και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, θα δούμε μερικές λεπτομέρειες συγκεκριμένες, αλλά σας έχω βάλει εδώ ένα κατάλογο ονομάτων πόλεων για να δείτε όσο ευρία είναι η επιλογή. Εγώ πήγα τελευταία στη Μασαλία και στην Προβυγγία γενικότερα για να δω ποιο ήταν το πρόγραμμα της πόλης αυτής, αλλά βλέπετε ότι έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των υποψηφίων πόλεων και των πόλεων που έχουν πάρει τον τίτλο της πολιτικής πρωτεύουσα Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξαν υποψήφιες και πόλεις από εκτός Ένωσης. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα εν συντομία τις αλλαγές. Γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως προς την επιτυχία ή μη των προγραμμάτων των πόλεων. Οι πόλεις βέβαια είναι τόσο διαφορετικές και τόσο πλούσιες σε κληρονομιά, ώστε είναι δύσκολο να δούμε τι θεωρείται ακριβώς επιτυχία. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένος τύπος. Εδώ βλέπουμε μία σειρά πόλεων όπου στην αρχή ήταν μόνο μεγάλες πόλεις, τώρα όλο και περισσότερο έχουμε και μικρότερες. Μερικές λιγότερο από 400.000 κατοίκους και από το 7 και μετά ιδίως είναι υποψήφιες και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις, τε, τεράστιοι συνοικισμοί. Μερικές φορές και ολόκληρες περιφέρειες. Υπάρχει λοιπόν μια νέα έννοια σήμερα περί του τι αποτελεί μια οικιστική Μητρόπολη. ας πούμε η Κωνσταντινούπολη από τις υποψήφιες μη ενωσιακές χώρες. Τώρα η χρηματοδότηση από τους τα ευρωπαϊκά όργανα και εκεί υπάρχει συνεχής αύξηση των χρημάτων που χορηγούνται στις πόλεις από λιγότερο από 200.000 ευρώ μέχρι 1,5 εκατομμύριο που είναι σήμερα η χρηματοδότηση. Και πάλι γρήγορα να σας πω ήταν, ποια ήταν τα κυριότερα επιτεύγματα. Οι πόλεις πώς υποβάλλουν υποψηφιότητα και πώς ορίζουν, καθορίζουν τους στόχους τους. Διαπιστώσαμε από το 5 και μετά ιδιαίτερα, στην τελευταία φάση θα έλεγα του προγράμματος, ότι η διαδικασία των προσφορών την χάνει πολύ περισσότερης προσοχής και από τα μέσα ήδη από την στιγμή που μια πόλη υποβάλλει την υποψηφιότητά της. Οπότε και είναι πολλές οι υποψήφιες βέβαια, όχι μόνο μία. Και γίνεται μια γενικότερη ανάλυση περί του τι είναι πολιτισμός και σε μερικές περιπτώσεις <clears throat> υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Το η Ισπανία και η Πολωνία υποβάλλουν υποψηφιότητες με πάνω από 16 πόλεις η καθεμία υποψήφιες. Στην Ιταλία ιδίως υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που θα μπορούσαν να γίνουν υποψήφιες και γι' αυτό πρέπει η διαδικασία επιλογής να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Το... Πρέπει το πρόγραμμα μιας πόλης να είναι καθεαυτού ενδιαφέρον και γίνεται και εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι κύριοι στόχοι είναι να αυξηθούν οι δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα και του πώς λειτουργεί σε αυτόν μία πόλη για να αποτελέσει καταλήτη οικονομικών εξελίξεων. Το κύριο θέμα είναι βέβαια να υπάρχει διαβούλευση μεταξύ όλων των οικονομικών και άλλων ενδιαφερομένων πολλοί θεσμοί δηλαδή να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα. Ε, βέβαια και η ποιότητα του ίδιου του καλλιτεχνικού προγράμματος έχει σημασία. Τώρα πώς μεταφράζεται αυτό σε πραγματική διαχείριση και εφαρμογή. Υπάρχει πολύ περισσότερη επαγγελματικότητα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Στην αρχή ήταν όλα αυτά πολύ κατακαιρματισμένα και πρόχειρα και τώρα ε, υπάρχει ένα προκαθορισμένο στυλ της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ε, κάποιο όραμα για την πόλη. Πολλές φορές γίνεται λόγος για αλλαγή της πόλης, προγράμματα από πολλούς και διαφορετικούς τομείς καθαρά πολιτιστικό αλλά και γενικότερης παιδείας, αθλητισμού, συνεργασία και πέρα από τις καθαρά τοπικές αρχές. Σημασία έχει επίσης ένα κεντρικό θέμα το οποίο να ενθαρρύνει ή να δίνει προτεραιότητες στην χρήση των διαθεσίμων πόρων και κάτι άλλο πολύ σημαντικό βέβαια να συμμετέχει ο κόσμος σε όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο πρότυπο, κάποιο μοντέλο που να εξηγεί και να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσφορές, πώς παρουσιάζεται το όραμα του προγράμματος, πώς γίνεται ο σχεδιασμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή ε, επειδή υπάρχουν πολλές μέθοδοι αποτίμησης και αξιολόγηση να τα συνδιασυνδέσουμε όλα αυτά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για θετικές επιπτώσεις αλλά δεν μπορούμε εύκολα να δούμε από την αρχή τι στοχεύει μια πόλη γιατί δεν προετοιμάζουν το πρόγραμμά τους με τόσο μεγάλη συνέπεια ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τι υπήρχε πριν και τι έγινε μετά ακριβώς. Υπάρχει ακόμη κάποιος κατακαιρματισμός. Εμείς πρέπει να καθορίσουμε ποια ήταν η πρόθεση και τι ακριβώς ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα υπάρχουν οι υποσχέσεις ή το όραμα των πόλεων και η πραγματοποίησή του. Πολλές φορές αυτό είναι φανερό γιατί στο Λίβερπουλ το 8, στο Τουρκού το 11 ε, είχαν υποβάλει προγράμματα που επέτρεπαν να γίνει αυτή η διασύνδεση εύκολα. Άλλα προγράμματα όμως δεν είναι τόσο σαφή. Να σας δείξω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει το πολιτιστικό πρόγραμμα μιας πολιτιστικής πρωτεύουσας. Πρώτον το καθαρά πολιτιστικό που είναι βέβαια καμιά φορά υποκειμενικό και άειλο αλλά είναι σαφές ότι μια πολιτιστική πρωτεύουσα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στις πολιτιστικές δραστηριότητες μιας πόλης. Στην δυνατότητα ας πούμε να ενισχυθούν ορισμένα δίκτυα, συνδυασμό, συνεννόηση παραγόντων με έναν κοινό σκοπό από το Λίβερπουλ μέχρι την Έσεν στο Ρουρ δημιουργούνται νέες συμμαχίες και συνεργασίες που επιβιώνουν και μετά το τέρμα, την περάτωση του πολιτιστικού προγράμματος της πρωτεύουσας. Ανοίγουν δυνατότητες για νέες συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικών χωρών αλλά και μεταξύ καλλιτεχνικών τομέων. Όπως σας είπα και πριν, καμιά φορά συνδέονται επιχειρήσεις με πολιτιστικό τομέα, με παιδεία γενικότερα. Υπάρχουν συνεργασίες με καινούργιες φιλίες. Νέο είδος συνεργασίας και εργασίας που μπορεί και αυτό να επιβιώσει μετά το πρόγραμμα, να λειτουργούν οι πόλεις δηλαδή διαφορετικά και να είναι πιο σημαντικός ο πολιτιστικός τομέας. Κάτι άλλο που είναι σαφές ότι μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις είναι ότι αλλάζει η εικόνα μιας πόλης. Και αυτό φάνηκε, είναι όλο και φανερότερο από τη στιγμή που επιλέχτηκαν ως πρωτεύουσες πόλεις που δεν ήταν προφανές να επιλεγούν ως τέτοιες ας πούμε η Γλασκόβη το 90 που είναι πόλη που έχει πολιτισμό αλλά έχει πολύ, είχε μέχρι τότε πολύ αρνητική εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοια παραδείγματα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Το Λίντς στην Αυστρία, ο Ισταβάνγκαρ στην Νορβηγία. Είναι πόλεις με γνωστή πολιτιστική δραστηριότητα αλλά όχι πολύ θετική εικόνα. και έτσι γίνεται και περισσότερος λόγος και συζήτηση για τις πόλεις αυτές και το πρόγραμμά τους. Και δημιουργείται βέβαια και περισσότερη δραστηριότητα στον καινούργιο αυτό κόσμο του ψηφιακ, τον ψηφιακό. Έχουμε μαζέψει πολλά στοιχεία από τις τελευταίες ιδίως εκδηλώσεις στο Τουρκού ας πούμε. Λοιπόν, χρειάζεται χρόνος για να εξηγήσουμε το πρωτογράφημα και βλέπετε σε πάνω από 7 χώρε ποιο είναι ο κύκλος των μέσων ενημέρωση. στα πλαίσια των προγραμμάτων πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στο έτος 0 βλέπουμε που η κάθε χώρα είχε πολιτιστική πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Βλέπουμε και πού είναι τα μέγιστα σημεία της κάλυψης στα μέσα ενημέρωση Εκεί όπου αυξάνεται η προσοχή πριν ή μετά τις εκδηλώσεις. Αυτό ε, συμπίπτει με τη διαδικασία υποβολής προσφορών υποψηφιωθήτων. Είναι η αρχή της διαδρομής εκεί. Τη στιγμή της συζήτησης, όχι τι συμβαίνει μόνο το γίνεται εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε από πλευράς πολιτιστικής και πώς όλα αυτά σχετίζονται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Από πλευράς ε, κοινωνικής, αυτό που συζητεί, τα αποτελέσματα που συζητούνται περισσότερο είναι τα αποτελέσματα στο πώς αντιλαμβάνεται η πόλη τον εαυτό της και η γειτονική περιοχή. Βλέπουμε πολλές πόλεις ισχυρίζονται ότι 50-90% τοπικού πληθυσμού αισθάνεται ότι η πόλη του είναι σε καλύτερη θέση αφού είχε τον τίτλο αυτό της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Είναι σημαντικές οι κοινωνικές συνέπειες φαίνεται κάτι υποκειμενικό και αυτό, αλλά η τοπική ε, περηφάνεια αυξάνεται και η στάση των τόπιων. Είχαν ε, περιοχές που έχουν οικονομικά προβλήματα και είχαν ειστερήσει οι πόλεις αυτές και είχαν περιθυροποιηθεί. Ε, μπορούν να περάσουν από ένα κομβικό σημείο όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος ε, βρίσκει ότι κάτι μπορεί να κάνει, ο πληθυσμό έχει κάποιο λόγο να μείνει. Κυρίως πανεπιστημιακές πόλει που μπορούν να προσελκύσουν φοιτητέ για να σπουδάσουν, αλλά έχουν πρόβλημα να του κρατήσουν. Αυτού του είδους λοιπόν οι πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν ένα λόγο ε, να πιστεύουν αυτοί τα πανεπιστήμια κλπ. Και, και οι φοιτητέ μάλλον ότι μπορούν να μείνουν. Άλλο κοινωνικό αποτέλεσμα. Βέβαια τα στοιχεία εκεί είναι πιο ανάμεικτα. Είναι η δυνατότητα να αυξηθεί αυξηθούν, να αυξηθεί το ακροατήριο και να, έχει, να είναι πιο ποικίλο το ακροατήριο. Ε, είναι πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να βρούμε αυτά αποτελέσματα, αλλά έχουμε ολόκληρη σειρά πόλεων από το Ελσίνκι το 2000, με την Κιμαράες και το Μαριγκόλ το 2012, που δείχνουν στοιχεία που δείχνουν ότι πάνω από το μισό του τοπικού πληθυσμού συμμετείχε στο πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο και αυτό λέει πολλά για την προστιθέμενη ε, αξία των δραστηριοτήτων. Δύσκολο να εξηγήσει κανεί τα γρήγορα αυτά που δίνουν τα στοιχεία όταν ολόκληρη σειρά γραφημάτων προσπαθούν να δώσουν μια εντύπωση τη όλη προόδου τη αλλαγή από το 85 μέχρι την πιο προσφατή ε, έκδοση. Με τα πιο προσφατά στοιχεία βλέπουμε το φάσμα των ε, του κόσμου, συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έτου, Αλλάζει αυτή η συμμετοχή. Περίπου ένα εκατομμύριο είναι οι παρουσίες σε κάποιες περιπτώσεις έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά που ξεχωρίζουν είναι το liverpool το 2008 και βλέπουμε ότι η πόλη αποφάσισε όχι μόνο να ασκήσει αυτές τις δραστηριότητε για ένα χρόνο, αλλά έχει τετραετές πρόγραμμα. 18 εκατομμύρια λοιπόν άνθρωποι μπόρεσαν άμεσα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους 9,8 εκατομμύρια συμμετείχαν, κοντά στα 10 εκατομμύρια που στις πιο πρόσφατες ε, τέτοιες ε, εκδηλώσεις ήταν ο μέσος όρος. Λοιπόν, κλείνοντας, άμεσα αποτελέσματα έχουμε λίγα στοιχεία όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κλπ. Είναι οι σχέσεις αίτιου και τιατούκι που είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Αλλά έχουμε ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά τη συνέπεια στον τουρισμό δηλαδή προσέλκυση τουριστών που αυτό επηρεάζει και την οικονομία των πόλεων. Έχουν πολλά στοιχεία για δραματική ανάπτυξη του τουρισμού κατά διάρκεια του έτους και τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι πόλεις μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 1, 2, 5 και μέχρι και 10 χρόνια μετά ε, του να είναι μια πόλη πολιτιστική πρωτεύουσα. Προσελκύει αυτή η πόλη περισσότερο κόσμο χάρη σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πιο περίπλοκο εδώ γράφημα που πρέπει να εξηγήσουμε τι δείχνει αυτή η γραφική παράσταση. Ότι η πιο κοινή τάση, έχουμε επιλέξει κάποιες πόλεις εδώ, πιο κοινό χαρακτηριστικό, βασικό σημείο, είναι το 100% παρουσιών στις εκδηλώσεις σε μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Και συνήθως βλέπουμε μια τάση ανάπτυξης οι παρουσίες αυξάνονται καθώς οδηγούμεθα προς το έτος αυτό και μετά μειώνεται. Και οι πόλεις ξαναλάζουν αυτή την τάση μερικά χρόνια αργότερα σε ξανά σε μεγαλύτερη ανάπτυξη να συμμετοχή εκδηλώσεις. Δύο με τρία χρόνια ε, χρειάζονται κάποιες χώρες, ε, κάποιες πόλεις συγγνώμη, για να αυξήσουν την τουριστική ροή. Σε κάποιες άλλες πόλεις μειώνεται απότομα τουρισμός άμα λήξει αυτή η περίοδος και σε άλλες πόλεις συνεχίζεται και πολλά χρόνια μετά τις εκδηλώσεις. Αυξάνεται και ο αριθμός των επισκεπτών ακόμα και μετά τη χρονιά που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα μια πόλη. Άρα οικονομικά αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προκλήσεις, προβλήματα. Ποια είναι. Έχουμε θετικές ειδήσει από τη μια πλευρά. Πολλές βασικές προκλήσεις που εντοπίστηκαν σε πρώτερες μελέτες, κυρίως αυτή του 94, και του Ράιτ του 2004, τα προβλήματα που είχαν εντοπίσει ξεπεράστηκαν. Είναι ασύνηθε να δει κανεί πόλει που δεν έχουν κάποια προσέγγιση για τη βιωσιμότητα και μισθωρική αναδρομή. Έχουν καλύτερη επικοινωνία οι πόλει και διάθεση του προϊόντο στην αγορά. Καλύπτονται οι διεθνεί ανάγκε. Υπάρχουν και άλλε προκλήσει. Όραμα. Να μην γίνει αντιληπτό ότι το πρόγραμμα αφορά μόνο μια ελίτ, αλλά όλους και χρειάζονται σωστά οικονομικά κοινωνικά προγράμματα. Και εδώ έχουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Σημαντικότατος στόχος και αυτός. Που ήταν πολύ περίπλοκος να αντιμετωπιστεί, να εξεταστεί και να παρουσιαστεί. Ο στόχος τώρα, η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, ποιος είναι. Από το 2005 είδαμε ότι είναι σαφέστεροι προσανατολισμοί υπάρχει καλύτερη υποστήριξη όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Οι πόλεις ακόμα παλεύουν να πετύχουν τα όσα έχουν ε, υποσχεθεί και για να πετύχουν. Γιατί, εν μέρη, το πρόγραμμα έγινε πάρα πολύ ελκυστικό για την τόπια οικονομία, για την κοινωνία. Και τα τοπικά προγράμματα επικρατούν. Θέλουν οι πόλεις ε, να αναλάβουν τι εκδηλώσεις για να προωθήσουν δικά τους προγράμματα. Και αυτό είναι βεβαίως σημαντικό καμιά φορά θεωρούν ότι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκή διάσταση είναι κάτι που πρέπει να κάνουν. Και τα μέσα ενημέρωση δεν αναφέρονται παρκώ στην ευρωπαϊκή ιδέα. Μιλάνε για την πολιτιστική πρωτεύουσα με τοπική απόχρωση κυρίω. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν υπέροχα προγράμματα που δείχνουν ότι δίνεται προστιθέμενη αξία όταν υπάρχει διασύνδεση με την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα προγράμματα ε, ε δεν έχουν δεν καλύπτουν τόσο καλά πλευρά στατιστική τη. Πρέπει να μετρήσεις ε, θεατές, αριθμό καλλιτεχνών που συμμετείχαν κλπ, δραστηριότητε και όταν κανείς συλλέξει και παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία ε, δεν βλέπει κανεί τόσο πολύ την ευρωπαϊκή διάσταση. Πρέπει να δείξουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση και προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται εκεί να δώσουμε ποιοτική διάσταση στα στοιχεία δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μόνο με γραφικέ παραστάσει. Και μετά η μεταφορά γνώση είναι το άλλο πρόβλημα. Πολύ δύσκολη σύγκριση, η προσαρμογή, η ανταλλαγή πληροφοριών. Για τα περισσότερα δίκτυα ήταν ανεπίσημα, θέμα γνωριμιών και συμπαθιών. Χρειάζεται πιο επίσημη προσέγγιση όσον αφορά αυτές τις ανταλλαγές για να είναι κάτι υποφελές για όλους. Από πλευράς λοιπόν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων δεν είναι πολύ καλή. Παρόλο που υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που μας δίνουν πολλά μαθήματα. Τώρα τα γενικά συμπεράσματα. Υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Μετά από τρεις δεκαετίες το πρόγραμμα έγινε ένα από τα πιο, πιο ορατές πρωτοβουλίες της με μεγάλο κύρος. Έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά. Αυτά μπορούν να αποδειχθούν εύκολα. Και σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν αποτελέσματα, ξεκινώντας από τη βάση ε, και μπορεί να αλλάξει η εικόνα της πόλης και της περιοχής. Για να ενισχυθούν τα προγράμματα πρέπει να συμβεί. Χρειάζεται σοβαρή προσέγγιση. Να, να υπάρχει ενθάρρυνση, να δοθούν συμβουλές, να υπάρχει σωστό όραμα, να εμπνέει το όραμα να τον στερνίζονται οι ντόπιοι, να έχει ευρωπαϊκή διάσταση, να αντιστοιχεί σε επιθυμίες των ανθρώπων, να μην είναι αποστασιοποιημένοι από το πρόγραμμα και τι εκδηλώσει Τι πρέπει να κάνουμε κι εμεί και οι πόλεις για να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού τομέα, γιατί είδαμε έναν κίνδυνο να υπάρχει τελευταία χρόνια, ότι το οικονομικό πρόγραμμα, ε, η οικονομική διάσταση είχε πάρα πολύ ισχυρή και καμιά φορά η πολιτιστική διάσταση κρυβόταν από κάτω. Άρα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με την οικονομία, με τους κοινωνικούς στόχους των πόλεων, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με σαφή προτεραιότητα που αφορά τον πολιτισμό. Χρειάζεται οι συμμετέχοντες αυτό να το καταλάβουν, ούτω ώστε να μην έχουμε σαν μοναδικό στόχο την προσέλκυση τουριστών, αποξενώνοντας διακριτικά στοιχεία της ντόπια κουλτούρας και χρειάζεται εξισορρόπηση σχέσεις μεταξύ πολιτικής στήριξης, ελέγχου και ανεξαρτησίας. Τα εξηγούμε αυτά λεπτομεράστερα στη μελέτη. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και η ομάδα. Αυτό το βλέπετε στην τελευταία διαφάνεια. Το μέλλον. Για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό είναι ένα τομέα όπου πραγματικά παραμένει ανοιχτή συζήτηση πολλά προβλήματα σχετίζονται με την προσπάθεια που έγινε από πόλεις που κάνουν προσπάθεια να δείξουν στους ντόπιου τι σημαίνει Ευρώπη. Ο κόσμος ήθελε αυτό να το καταλάβει και να το καθορίσει μόνος του. Είναι σημαντικό λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό, οι πολίτες να μην θεωρούν ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ ντόπια και ευρωπαϊκής διάστασης εφόσον είναι Ευρωπαίοι ελώστε και αυτό που είναι τοπικού ενδιαφέροντος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ευρώπης. Και αν πρέπει με διαφορετικό τρόπο να το καθορίσουν αυτοί, αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα έχει γίνει πάρα πολύ ελκυστικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον και την χάνει μεγάλη προσοχή από τα ΜΜΕ. Και είναι σημαντικό και βοηθά την ευρωπαϊκή συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα. Όταν υπάρχουν συζητήσει, διασκέψει, σεμινάρια, εργαστήρια, ξεκινάει ο διάλογο. Και η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Για μεταφορά γνώση για το μέλλον. Χρειαζόμαστε καλύτερο επίσημο πλαίσιο. Τυποποίηση για τη συλλογή των στοιχείων. Θέλουμε βασικούς δείκτες κλειδιά, λίγου, για να συλλέγουν στοιχεία με παρόμοιο τρόπο οι πόλεις για να υπάρχει συγκρισιμότητα στοιχείων. Όχι μέχρι τώρα γιατί αντιμετωπίσαν πολλά προβλήματα για τη συλλογή στοιχείων για τη μελέτη. Και υπήρχαν προβλήματα συγκρισιμότητας και ποιότητας. Αυτά και περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. I have a lot of uh, Έχω πολλές ερωτήσεις. Ε, και μετά ο Σάντρος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πραγματικά την κυρία Γκαρθία για αυτήν την ε, ιδιαίτερα σαφή, πλήρη παρουσίαση που τεκμηριώνει θέματα ε, απόψεις που βέβαια ήδη είχαμε αλλά ακριβώς τις ε, θεμελιώνει. Η πρωτοβουλία αυτή όντως ε, έχει προστιθέμενη αξία και επειδή τώρα είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία, είναι σημαντικό να καταδείξουμε ότι οι πρωτοβουλίες μας προσφέρουν προς τη θέμα αξία για τους πολίτες, για τις πολιτικές μας. Αποδείξατε ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις αλλά και σε ακτινοβολία. Ξέρουμε ότι το πιο δύσκολο είναι πάντα να αποτιμήσει κανείς τις επιπτώσεις πού ακριβώς είναι και πώς η προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μας δώσατε στοιχεία αριθμητικά, πολύ εύγλωτα, ως Γαλλίδα Ευρωβουλευτής. Τον Σεπτέμβριο, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας, πέρα από την ε, αντιπροσωπεία, την επίσημη, πήγα στη Μασαλία για να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε τι επιπτώσεις έχει στην ε, αστική ανάπτυξη. Έχουμε μία διαπολιτική ομάδα για την ε, αστική ανάπτυξη ακριβώς. Είχαμε επιλέξει ως στόχο Μασαλία ε, και Προβυγγία 2013. Είδαμε ότι δημιούργησε δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων και της υπαίθρου Δώσατε το στοιχείο 600 εκατομμύρια επενδύσεων, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερες οι επενδύσεις και θα έχουμε 8 εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι το τέλος του χρόνου και κάποιες άλλες διαπιστώσεις που κάναμε το Σεπτέμβριο. Πρώτα απ' όλα παίζει καταλητικό ρόλο αυτός ο τίτλος Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα έχει οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Διαπιστώσαμε ότι οι Μαρσεγέζοι μπόρεσαν να ξανακερδίσουν την πόλη τους, άλλαξαν την εντύπωση που έχουν οι ίδιοι για την πόλη τους. Από την αρχή του 2013 υπόθηκαν πολύ θετικά στα μέσα για τη Μασαλία, συγγνώμη, προηγουμένως λέγονται αρνητικά για την εγκληματικότητα, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ε, μαφία κτλ. Αλλά ναι, μεν δεν υπήρξε βέβαια στην αρχή πολύ ενδιαφέρον για την Μασαλία ω πολιτιστική πρωτεύουσα, γιατί λόγω τη αρνητική εικόνα θεωρούσαν ότι θα αποτύχουν. Είχαν πάει τον Ιανουάριο για την ε, έναρξη και έκτοτε ε, να σα δώσω μερικά παραδείγματα του ρόλου του καταλητικού που αναφέρατε και που είναι αλήθεια. Μία πρωτοβουλία για ένα μουσείο μπόρεσε να ξεκινήσει λόγω ακριβώς ε, αυτής της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Έτσι έδωσε και το γαλλικό κράτος ε, κονδύλια. Το κράτος μάλιστα το είχε πει ότι αν γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα θα χρηματοδοτήσουμε το μουσείο. Έγινε λοιπόν αυτό. Πολύ θετικό. Και όλες οι ανακαινήσεις κτηρίων ε, στο λιμάνι της Μασαλίας, το οποίο είχε υποβαθμιστεί πολύ, το Σιλό, για παράδειγμα, είναι θέατρο που έγινε σε μια παλιά αποθήκη στο λιμάνι και επίσης και ιδιωτικές επενδύσεις για ένα Intercontinental πέντε αστέρων όπου πηγαίνουν υψηλού επίπεδου πελάτες και από διάφορες συνοικίες όπου είχαν κατέβει άνθρωποι σε διαδηλώσεις είδαμε σε αυτές τις διάφορες γειτονιές έγιναν αλλαγές μακροπρόθεσμες λοιπόν και φυσικά οι υποδομές θα μείνουν, άλλαξε η εικόνα της πόλης. Και φυσικά ε, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των επισκεπτών για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και κάποιες επενδύσεις στο λιμάνι που ποτέ δεν θα είχαν γίνει εάν δεν είχε αποδοθεί αυτός ο τίτλος. Επιτύχαμε λοιπόν τους στόχους μιας, ευρωπαϊκής, μιας ε, ανάπτυξης ε, ευφυούς και χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, ε, αυτά που είπατε, επίσης για τη μεταφορά γνώσεων και είμαστε περισσότερο σε μια ευρωπαϊκή διάσταση, όχι απλώς σε ένα πρόγραμμα, όχι να είναι κατάλογος όπως τα πείματα του Πρεβέρ. Πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ της τοπικής και της ευρωπαϊκής διάστασης και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Γίνονται επενδύσεις. Διαπιστώσαμε γιατί πήγαμε για να δούμε και την ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Είδαμε επενδύσεις και από το Περιφερειακό Ταμείο και από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Υπάρχει λοιπόν ε, συνεργασία λόγω από τη μία του τίτλου πολιτιστική πρωτεύουσα και των άλλων δυνατοτήτων που παραγνωρίζονται πολλές φορές αλλά που αναβαθμίζονται μέσω αυτού του τίτλου. Φυσικά λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε βελτιώνοντας αλλά νομίζω ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος ε, σε τρεις δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής μας, Κορέα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ την δόκτωρα Γκαρσία διότι η παρουσίασή της και αυτά που μας παρουσίασε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ακριβέστατα, επίκαιρα και χαίρομαι που κάποια σημεία που υπογράμμισε εμπεριέχονται στην έκθεση που υθέτησε το Κοινοβούλιο, το ενέκρινε η Επιτροπή μας. Εργαζόμαστε καλά λοιπόν, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ένα από τα τελευταία πράγματα που είπατε μου έκανε εντύπωση η σχέση μεταξύ πολιτών και κάποιων πόλεων με την ευρωπαϊκή διάσταση. Δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούμε να βρούμε σχέση τοπικών πτυχών με γενικότερες πτυχές. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Να ζητήσω κάτι. Όταν κάναμε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο, Μεταξύ των θεμάτων που συζητήσαμε εμπεριείχονται δύο πτυχές επί των οποίων ήταν πιο εχθρικό το Συμβούλιο και αντιμετώπιζε δυσκολίες να δεχτεί τις παρατηρήσεις μας. Και ένα από αυτά τα σημεία ήταν η Ευρωπαϊκή Διάσταση. Στο τέλος δέχτηκε αυτό το σημείο. Μετά υπήρχε πρόβλημα όμως όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας που υπογραμμίζουμε εμείς σαν ένας από στόχους, σαν έναν από τους στόχους του προγράμματος της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης και ένα από τα μέσα που θα μπορούσε ε, θα μπορούσε να χρησιμεύσει αμέσω μάλλον. Βάσει της μελέτης και της εμπειρίας, τι έχει να πει η δόκτωρ όσον αφορά τις αναλύσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ Μάρκο. Η κυρία Τρίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστώ την κυρία Γκαρσία. Αναφερθήκατε στο δίκτυο των ε, πολιτιστικών πρωτευουσών. Ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των πόλεων ε, και υπήρχαν θετικά αποτελέσματα και είναι ανεπίσημο δίκτυο μέχρι τώρα. Και μιλήσατε για την επισημοποίηση της μεταφοράς γνώσης. Θα μπορούσατε να συστήσετε κάτι Θέλετε αυτά τα δίκτυα να επισημοποιηθούν, να είναι πιο επίσημο το πλαίσιο. Ε, υπάρχουν στοιχεία μετά ότι μετά το έτος ε, των εκδηλώσεων υπάρχει μια βιώσιμη υποστήριξη το, του πολιτισμού στις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Είναι μεγαλύτερη στήριξη από ό,τι κατά παρελθόν ή δεν υπάρχουν πλέον χρήματα και δεν μπορεί να συνεχιστεί η στήριξη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και θέλω να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις σας. Αυτά που είπε η επίσης, δηλαδή να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και ποιες είναι οι δυσκολίες. μείωσα αυτά που είπατε. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν οι πρωτεύουσες, οι πόλεις να χρησιμοποιήσουν την ιδέα αυτή της πολιτιστικής πρωτεύουσα για να προωθούν τοπικά θέματα και ότι δεν προωθείται παρκώς η ευρωπαϊκή ιδέα. Δεν το καταφέρουν αυτό οι πόλεις, είπατε. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι δεν μπορεί να αποχρεώσει κανείς τους πολίτες να το κάνουν αυτό και σωστά είπατε ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις ε, για το πώς μπορεί να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση. Κάποιες πόλεις λησμόνησαν αυτή τη διάσταση από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Πώς θα πετύχουμε να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση. Δεύτερον, κάποιες από τις επόμενες πόλεις θεωρείτε θα το καταφέρουν αυτό. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Με το όρχους είδαμε ότι προσπαθεί, θα προσπαθήσει η πόλη να ξεκινήσει από την ευρωπαϊκή διάσταση. Δηλαδή να μην εξετάσει το όρχους, τι θα κάνει η Ευρώπη για το όρχους, αλλά τι θα κάνει το όρχους για την Ευρώπη. Ίσως πρέπει να αλλάξει η στόχευση. Όταν υποβάλλουν υποψηφιότητα οι πόλεις να είναι πολιτιστικές πρωτεύουσε. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν θέλετε οι πόλεις να προσπαθήσουν να συζητούν το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας πρέπει ήδη να βλέπετε πώς παρουσιάζουν τα προγράμματα τους και κατά πόσο θα συμπεριλαμβάνεται αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση. Έχετε κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Ο Σαντιάγο Φίσας. Ευχαριστώ και συγχαίρω και την εισηγήτρια για τη θαυμάσια εκθεσή της. Δύο σχόλια, παύλα ερωτήσει. Πρώτον. Η τοπική κουλτούρα. Και εγώ ήμουν στη Μασαλία, προέδρευα σε μια συνεδρίαση, μάλλον μια επίσκεψη θα έλεγα. Ήταν και ο Μάρκος Χορέα και άλλοι συνάδελφοι. Το πρόβλημα που διαπιστώσαμε, το μόνο παράπονο, μιλώντας και με τους ε, ανθρώπους εκεί μας έλεγαν όλα είναι θαυμάσια έγιναν πολλά πράγματα έγινε αυτό το μουζέμ όλα αυτά που είπε η συνάδελφος αλλά, αλλά, αλλά τι γίνεται με τον τοπικό πολιτισμό τα χρήματα που συνήθως δίνονται για τοπικές πρωτοβουλίες για τη ζωή του τοπικού πολιτισμού δίδονται για αυτή την ε, εκδήλωση μεγάλης έκτασης και αυτό είναι κρίμα όχι μόνο για τη Μασαλία αλλά και γενικότερα. Ισχύει για όλε τι ε, πολιτιστικέ πρωτεύουσε, Κάτι άλλο ε, που έχει να κάνει με αυτό, που, είπε η κυρία Τρίπελ. Τι θα γίνει μετά. Πολύ σημαντικό. Όχι μόνο θα πρέπει να βοηθήσει κατά τη διάρκεια τη πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά θα πρέπει να μεταμορφώσει όλη την πόλη, να αφήσει ε, βεβαίω μεγάλε εγκαταστάσει. αλλά πρέπει να δούμε ότι στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του τίτλου Αναφέρεται επίσης ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μετά την πρωτεύουσα. Στο μέλλον δηλαδή. Ευχαριστώ. Από πλευράς μου. Ε, από ό,τι μπορούσα να ακούσω γιατί με συγχωρείτε καθυστέρησα μπορώ να σας πω ότι θεωρώ πολύ πιστικά αυτά τα οποία άκουσα. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, ομιλήτρια. Όμως θα σας μιλήσω τώρα για τη δική μου πείρα από την δική μου χώρα και να αναφέρω τρία παραδείγματα. Ε, από τις πόλεις Σιμπιού, Ερμανστάτ, δύο πόλεις λοιπόν της Ρουμανίας αλλά θα μπορούσα να αναφέρω και την Πέτς, την πόλη Πέτς της Ουγγαρίας και το Κόζιτσε της Σλοβακίας. Κοσόν το λέμε ουγγρικά. Πήγα σε όλες αυτές τις πόλεις και διαπίστωσα, τι διαπίστωσα λοιπόν. Συνέβαλε ιδιαίτερα η πρωτοβουλία αυτή ε, στην ανάπτυξη των πόλεων. Αυτές ήταν πόλεις που ανήκαν στην Αυστρογγρική Αυτοκρατορία. Αυτός ο τίτλος λοιπόν της πολιτιστικής πρωτεύουσα είχε ε, τρομερή επίπτωση σε αυτές τις πρώην χώρες. Ο τίτλος αυτός, η ετικέτα αυτή λοιπόν, ε, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, επέτρεψε την ανάπτυξη των πόλεων αυτών. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που βοηθάει πολύ τις χώρες αυτές, τις πόλεις αυτές, Είναι ένας τίτλος λοιπόν που επιτρέπει σε αυτές τις πόλεις να ενταχθούν καλύτερα στην Ένωση. Ο τίτλος αυτός επιτρέπει στις πόλεις να αναπτυχθούν αλλά και στις μικροπεριφέρειες γύρω τους, στην εδώ χώρα τους δηλαδή. Βεβαίως έτσι εντάσσονται καλύτερα οι πόλεις. Επιτρέπει και την αλληλοκατανόηση μεταξύ πόλεων. Οι πόλεις ε, αλλά και οι εθνότητες, οι μειονότητες, ε, οι θρησκείες ε, μπορούν να αλληλοκατανοηθούν καλύτερα. Το Σιμπιού είναι μια πόλη Είναι λοιπόν μια πόλη όπου υπάρχουν πολλές μειονότητε. Και αυτό ισχύει και για το Κόζιτσε, το Κοσάρ στα Ουγγρικά. Και για την ε, θαυμάσια πόλη του Πέτς και στην Αυστρία. Στην Αυστρία υπάρχουν πολλές πόλεις ε, που έχουν μειονότητες όπου υπάρχει παρουσία της ιστορίας τους πολύ έντονη. Μια ιστορία με πολλές ε, διαστάσεις. Υπήρξε λοιπόν μια διαδικασία συμφιλίωσης και στο ΣΥΜΠΙΟΥ. Στο ΣΥΜΠΙΟΥ υπάρχει ένα ε, λουθυρανικό πολιτιστικό κέντρο ε, το οποίο ε, κυρίως ήταν για την σαξονική κοινότητα. Γιατί θυμάστε ότι ήταν, όπως είπα, στην Αυστρογγλική Αυτοκρατορία και η πόλη αυτή. Βοήθησε λοιπόν μέσω του πολιτισμού την προσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων. Είναι η απόδειξη ότι βοηθάει. Είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η πρωτοβουλία. Γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε και η Τιμισοάρα, Τέμεσοάρα στα Ουγγρικά, όπου ξεκίνησε η επανάσταση, ξέρετε, για τη Ρουμανία. Ήμουν και εγώ παρόν. Με είχε συλλάβει πριν από 24 χρόνια το καθεστώς ε, Τσαουσέσκου στην Τιμισοάρα υπήρξε εξέγερση ε, μεταξύ 10, στην οποία συμμετείχαν 10 διαφορετικές ε, μειονότητες, κοινότητες, θρησκευτικέ κοινότητες. Ενωμένοι εξεγερθήκαμε και μπορώ να σας πω η μισοάρα είναι ε, αυτή τη στιγμή υποψήφια για τον τίτλο της πολιτικής πρωτεύουσα. Θα μπορούσα να φέρω και το Κλούζνα Πόκα. Κλάουζενμπόγκ είναι το παλιό του όνομα. Ή Κόλος Βάρτο λέμε ουγγρικά. Ε, και η πόλη Σιουκίλ η Καϊφέλ στα Ουγγρικά και επίση και αυτή είναι υποψήφια και θα ήμουν ιδιαίτερα θετικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει και αυτές τις ε, πόλεις στη χώρα μου συνολικότερα. Επίσης σας ευχαριστώ άλλη μια φορά και καταλήγοντας να τονίσω κάτι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή αλλά και η εθνική και η τοπική διάσταση πρέπει όλες να είναι παρούσες. Αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σον Κέλλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια στη δόκτωρα Γκαρσία για την παρουσίασή της. Σημειώνω επίσης ότι λαμβάνει υπόψη τη σοβαρά τις παρατηρήσεις μας και αυτό είναι πολύ θετικό. Μερικά σχόλια. Πρώτον, σημειώθηκε καμία σοβαρή αλλαγή στη στάση, στην νοοτροπία των πολιτών στις πολιτιστικές πρωτεύουσες ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δηλαδή λιγότερος ευρωσκεπτικισμός μετά τα προγράμματα αυτά και περισσότερος ευρωπαϊκός ενθουσιασμός. Δεύτερον, στην παρουσίασή σας σημείωσα ότι οι διαφορές πόλεις έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, βέβαια αυτό είναι φυσικό, αλλά ιδιαίτερα τι κληρονομιά αφήνουν οι περίοδοι πολιτιστικής πρωτεύουσας. Είπατε ότι σε τοποθεσίες πόλης, αυξάνεται ο τουρισμός, σε άλλες μειώνεται. Με αυτή τη βάση λοιπόν, σε αυτή τη βάση. Τι προτείνετε για τις πόλεις στο μέλλον ώστε να συνεχίσουν να ωφελούνται από τα προγράμματα πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Στην αρχή της συζήτησης είπα ότι μαζί με τον εισηγητή θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με την αστική ανάπτυξη. Ότι πρέπει να είναι ένας από τους στόχους. Αλλά δεν το διαπίστωσα καθόλου σε αυτά που είπατε. Βλέπω ότι κάπου αναφέρεστε στην εικόνα των πόλεων. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με την αστική ανάπτυξη. Θα ήθελα το κείμενο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο των πολιτιστικών πρωτευουσών, ούτω ώστε να υπάρξει, όφελη, να υπάρξει ο, όφελος, για παράδειγμα, για τις ε, ε, παλιές ε, βιομηχανικές περιοχές ε, που τώρα είναι σε παρακμή και για τις ε, υποβαθμισμένες ε, περιοχές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πολιτιστικούς σκοπούς. Αυτά υπάρχουν πολύ στο Λίβερπουλ. Στις συζητήσεις με το Κορεπέρ θα μας βοηθούσε πολύ αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν μόνο δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες που επιχείρησαν η ενδοχώρα να συμπεριληφθεί το Λουξεμβούργο ε, επειδή ήταν για δεύτερη φορά πολιτική πρωτεύουσα, θέλησε να αξιοποιήσει και το Grund. Δηλαδή είπε να βοηθήσει και την ευρύτερη περιοχή Μοζέλας, ε, Ρινανία Παλατινάτο, ε, Λουξεμβούργο του Βελγίου. Πολύ καλό αυτό. Και αυτό θα έπρεπε να τονιστεί περισσότερο. Διότι μια πόλη από μόνη της είναι πολύ μεμονωμένο. Πρέπει και ενδοχώρα η περιοχή γύρω τα περίχωρα να συμπεριληφθούν. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κάνουμε τεράστια εργασία για να πιέσουμε και να πείσουμε την Κομισιόν. Στην αρχή η Κομισιόν ήταν πολύ αρνητική, εν μέρη ίσως έχει μεταπιστεί, δεν ξέρω αν είναι παρούσα εδώ για να μας πει. Α, είναι παρούσα, ωραία, άρα μπορεί να μας πει. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει μου. Να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Α, όχι, πρώτα η Δόκτωρ Γκαρσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Καλό να ξεκινήσω από την τελευταία. Το θέμα της αστικής ανάπτυξης θεωρούσα ότι θα μπορούσε να επανέλθει στη συζήτηση. Στη βασική μελέτη βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα τμήματα. Εξετάζουμε τον πραγματικό αντίκτυπο, φυσική διάσταση, ποια στοιχεία υπάρχουν, ποια δεν υπάρχουν για την προστιθέμενη αξία, του συσχετισμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσα και των διαφόρων εκδηλώσεων με πραγματικές εξελίξεις. Και τι είδαμε, ότι πολλές πόλεις χρησιμοποίησαν τις πρωτοβουλίες και τις διασύνδεσαν με δικά τους προγράμματα για αστική ανάπτυξη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Έλαβαν υπόψη δηλαδή την ανάπτυξη, τη φυσική ανάπτυξη των υποδομών όπως για τη Μασαλία, όπως με το Λίβερπουλ. Δηλαδή το άνοιγμα της πόλης προς τις υδάτινες εκτάσεις. Η αστική ανάπτυξη πρέπει να γίνει αντεληπτή σε πολλές διαστάσεις. Έχουμε φυσική διάσταση, θέμα κατασκευών οικοδομών, μεταφορές, διασυνδέσεις, διασυνδέσεις γειτονιών, πώς εξασφαλίζεις το ότι αυτά τα προγράμματα βοηθούν την διασύνδεση, εκ νέου διασύνδεση διαφόρων γειτονιών που έχουν απομονωθεί και που δεν συνδεόταν με το κέντρο της πόλης. Και τι είδαμε. Αντιφατικά στοιχεία υπάρχουν γι' αυτό. Έχουμε παραδείγματα πολύ θετικών αποτελεσμάτων, σαφών αποτελεσμάτων, με επενδύσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα, όπου υπάρχει σωστή χρηματοδότηση και στήριξη του προγράμματος και εκεί έχουμε τα πιο απτά αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα για πολλούς στο Λίβερπουλ και το ίδιο θα συμβεί και στη Μασαλία. Η χρονιά της πολιτιστικής πρωτεύουσα ε, σήμαινε για το Λίβερπουλ ότι άνοιξε ένα νέο εμπορικό κέντρο. Κάτι πολύ ορατό σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα νέο κέντρο συνεδριάσεων. Και τώρα μπορεί να οργανώνται εκεί διάφορες συναυλίες και διασκέψεις στην πολιτική Και για τη Μασαλία θα ανοίξει το μουσείο και θα αναπτυχθεί περιοχή. Αυτά είναι υπέροχα. Σε κάποιες περιπτώσεις, άλλα παραδείγματα που αναφέρονται και στη μελέτη, βλέπουμε πόλεις που είχαν επενδύσει πολύ στη φυσική ανάπτυξη αλλά δεν είχαν σαφές πρόγραμμα για συνέχιση και είχαμε τελικά αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέπουμε μία αποδοχή ότι η διάσταση της αστικής ανάπτυξης είναι σημαντικότατη και άκρος επωφελής όταν υπάρχει διασύνδεση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και με τις ιδιαιτερότητες της χρονιάς συγκεκριμένη της πολιτιστικής πρωτεύουσα και μπορεί να πετύχεις αποτελέσματα σωστά με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά όχι αν τα κάνεις όλα βιαστικά. Τα καλύτερα αποτελέσματα είναι τα παραδείγματα αυτά που λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες περιοχές της πόλης, διάφορες γειτονιές και εφαρμόζονται διάφορα μικρότερα προγράμματα που δεν φαίνονται στις γραφικές παραστάσεις. Τώρα, πώς να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε εχθρική στάση του Συμβουλίου στον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση και πώς μπορούμε να συζητήσουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ποια μέσα υπάρχουν που θα μας βοηθήσουν, το είπε ο κ. Σκουρή αυτό. Πρέπει να θυμηθούμε κάτι. Για κάθε πόλη και κυρίως την πολιτιστική πρωτεύουσα η Ευρώπη σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για το Λίβερπουλ βλέπουν πιο πολύ που στον Ατλαντικό στο Λίβερπουλ. παρά με την υπηρετική. Δεν κοιτούν τόσο πολύ που στην υπηρετική Ευρώπη. Άρα διασυνδέσουμε το Μανχάταν με τη Νέα Υόρκη και με την Σανγκάη και με την ε, κινέζικη κοινότητα. Για να δουν την ευρωπαϊκή διάσταση ε, θα έπρεπε να υπάρχει διασύνδεση και με αυτές τις κοινότητες. Η ευρωπαϊκή ιδέα και σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και με τις άλλες υπήρους, με τη ΣΥΠΑ, με την ε, Ασία στην περίπτωση μας είναι η σχέση με την Βόρεια Αφρική. Περίπλοκο, περίπλοκη εικόνα, περίπλοκο μοσαϊκό. Μιλάμε για σύμβολα και πώς μεταφράζονται στην έννοια της ταυτότητας που να μπορεί να συνοψιστεί. Είναι κάτι εύκολο, όχι δεν είναι εύκολο να συνοψιστεί. Και αυτή είναι η ομορφιά του έτους αντί να έχουμε ε, εκδηλώσεις για κάποιες εβδομάδες. είναι καλές οι συζητήσεις για αυτό το θέμα. Κάποιος μπορεί να πει εγώ είμαι Ευρωπαίος αλλά η πρόγονή μου είναι από την Κίνα αλλά ζω αρκετά χρόνια εδώ και αυτό πρέπει να συζητείτε. Για κάποιες κοινότητες λοιπόν το συνέστημα ότι κάτι είναι άσχετο με μας αφήνεται σε προκαταλήψεις. Δηλαδή στο πώς καθορίζουν ε, την, ε, την Ευρώπη και κατά πόσο η ιστορία του σχετίζεται με την Ευρώπη. Και γι' αυτό βοηθά το ότι διαρκεί ένα χρόνο η όλη διαδικασία. Στο μέλλον θα πετύχουμε καλύτερα πράγματα αν ενθαρρύνουμε τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τον περίπλοκο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής διάστασης και να δεχθούν ότι ίσως η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες εκδηλώσεις με σημαντικές προσωπικότητες, αστέρια από την Ευρώπη που αστορκήσουν τους τουρίστες αλλά ίσως για τους ντόπιου χρειάζεται εκδήλωση, ε, χρειάζονται εκδηλώσεις τοπικού επίπεδου, να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι είναι πιο υπερήφανοι για τι εκδηλώσει του, ενδιαφέρουν περισσότερο, λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση εκδηλώσει τοπικέ. Και απαντώντα σε ένα άλλο ερώτημα, δηλαδή αν υπάρχουν στοιχεία το ότι το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα αλλάζει τον κόσμο που αντιλαμβάνεται ο κόσμος στην Ευρώπη ή σκέφτονται περισσότερο οι άνθρωποι την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουν πολλές προκαταλήψεις. Κυρίως όταν μιλάμε για ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, εκεί υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Κάποιες χώρες είναι πιο ενθουσιώδεις για ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες, κυρίως τα τελευταία χρόνια, ε, ίσως έχουν προβλήματα με αυτή την ιδέα. Άρα είναι θέμα προκαταλήψεων και διαφόρων συσχετισμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κάποιες πόλεις και κάποιες κοινότητες θα αισθανόταν πιο υπερήφανες αν μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα. Να, να, να πούν γιατί αισθάνονται αποσυνδεδεμένες οι κοινότητες από την Ευρώπη και ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια πια είναι ότι στα βασικά προγράμματα δεν βλέπουμε τι γίνεται όσον αφορά την πρόθεση των προγραμμάτων, όμω πολλέ πόλεις, πολιτιστικέ πρωτεύουσε που έχουν πανεπιστήμια κυρίω, πολύ συχνά ε, οργανώνουν συζητήσει μεταξύ των φοιτητών, εφαρμόζουν προγράμματα σε τοπικό επίπεδο και πολύ συχνά ε, συζητείται αυτό. Τι σημαίνει αυτό για μας, πόσο το αποτιμούμε, τι σημασία έχει για μας. Μπορεί να συμβεί αυτό σε τοπικό επίπεδο. Καμιά φορά όταν δεν είναι πρωτοσέλιδο η εκδήλωση, σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωση αντιμετώπισαν πιο διαφορετικά το, την εκδήλωση, πιο αρνητικά, ε, το θέμα πιο αρνητικά. Οι άλλε φορέ υπάρχουν άλλα προβλήματα. Χρειάζεται δουλειά για τη σωστή αντιμετώπιση και προβολή. Χρειάζεται ποιοτική αξιολόγηση. Μπορούμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για πολύ μικρά προγράμματα που έκαναν τη διαφορά. Σας ενθαρρύνω εσάς να δείτε πρωτοβουλίες. Όπως η πόλη στο περιθώριο στην άκρη, ε, ε όπως είναι Λίβερπουλ, διασύνδεση του Λίβερπουλ με τη Μασαλία, με την Νάπολη, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα αντιμετωπίζονται δύσκολα προβλήματα, προβλήματα εγκληματικότητα, βία σε διάφορε πόλει, που αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο τη Ευρώπη αυτέ οι πόλει. Αλλά ταυτόχρονα αυτέ οι πόλει έχουν πολύ ισχυρή δημιουργική και πολιτιστική βάση και έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσε ζητήσει σε αυτό το πλαίσιο που δυστυχώ δεν προευλήθησαν επαρκώ τα ΜΜΕ και δεν προβλήθηκαν και δεν μπήκαν στα πρωτοσέλιδα αυτές οι εκδηλώσεις. Με τα χαράς να συνεχίσω τη συζήτηση Προσπαθώ να δω δύο-τρία άλλα σημεία που είχαν θυγεί. Το θέμα της κοινωνικής συμμετοχής και πώς οι πολίτες κατά πόσο αισθάνονται ότι οι εκδηλώσεις τους αφορούν. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται. Όταν μιλάμε για πολιτιστικά θέματα υπάρχουν πολλές αντιλήψεις περί αυτού. Και εδώ δεν μιλάμε για καλλιτεχνικέ εκδηλώσει. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα δεν είναι το ίδιο σαν ένα φεστιβάλ. Είναι μια δυνατότητα μια πόλη να προβληματιστεί, να εξετάσει τον εαυτό της, στις διάφορες πτυχές, κάποιες πόλεις το κάνουν διασυνδεόμενες με θρησκεία, μαθητισμό κλπ. Και κάτι πολύ ευρύτερο, πολύ ευρύτερο πλαίσιο από ότι απλώς οι καλές τέχνες και η τέχνη γενικά. Άρα χρειάζεται δραστηριότητα σε πολλαπλά επίπεδα. Οι οικονομικοί στόχοι, προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών. Σημαίνει ότι οι πόλεις θέλουν να έχουν πρωτοβουλίες που προβάλλονται να έχουν μεγάλα μπαλέτα, να, όπερες κλπ. Και αυτά ίσως να μην αφορούν οι εκδηλώσεις στην τοπική κοινότητα. Στη Μασαλία το είδαμε. Τι γίνεται στο κέντρο της πόλης, με τις κοινότητες του κέντρου της πόλης. Δεν ξέρω πόσο θα ενδιαφερόταν αυτοί οι άνθρωποι για το μουσείο. Αν και καλά τα πάει το μουσείο σαν δημόσιος χώρος για όλους. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα άλλα κοινωνικά προγράμματα που δεν ενδιαφέρουν τα μέσα ενημέρωσης και τους επισκέπτες. Και όπως είπα έχουν αυξηθεί αυτά, υπάρχουν. Ε, πολύ συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανακοινοθέντα τύπου, ούτε στα φυλάδια που θα σας στείλουν, αλλά όλο και περισσότερο εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα στο τοπικό επίπεδο. Μεγάλη πρόκληση ποια είναι. Αν κάνετε μια έρευνα και ρωτήσετε, βολιδοσκόπηση και ρωτήσετε του πολίτε τι θυμόσαστε για την πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη, τι είχε αξία για εσά. Κάποιοι θα σα πούν ίσω ότι του άρεσε κάτι πάρα πολύ και λυπούνται που η ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα δεν αφορούσε αυτό και το πρόγραμμα ήταν μέρος αυτού αλλά δεν είχε προωθηθεί σε κάτι τέτοιο. Άρα έχουμε και θέμα του πώς παρουσιάζουμε τις εκδηλώσεις και πώς σχετίζονται με μια εκδήλωση οι άνθρωποι. Να μην θεωρούν ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στα μουσεία και στα θέατρα αλλά και αλλού. Γίνεται δουλειά και στους δρόμους και στις γειτονιές. Όλο και περισσότερο συμβαίνουν αυτά, σε τοπικό επίπεδο εκδηλώσει δηλαδή, και τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά πολλές φορές και μεταμορφώνται κοινότητε. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό θα πρέπει να ε, προωθηθεί και να συμπεριληφθεί στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Και κάτι άλλο υπόθηκε, κάτι διαφορετικό στο οποίο ήθελα να απαντήσω, επενδύσεις. Κάποιες πόλεις ναι, κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή, πώς σχετίζονται αυτοί αυτές οι πτυχές με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Όταν αξιολογούμε την επιτυχία η την αποτυχία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη μακροπρόθεσμη σκοπιά. Μια πόλη που εξέτασα προσεκτικότατα ήταν η Γλασκόβη το 90. Αν γινόταν η μελέτη 95-96 θα θεωρούσε κανεί ότι ήταν αποτυχία. Το 2000, 2002, 2003 κλπ. μετά από 10 χρόνια βλέπει κανείς ότι έχει γίνει όλος ο κύκλος και μπορεί να δει κανείς πραγματικά τα αποτελέσματα θαυμάσια, υπέροχη μεταμόρφωση της πόλης έλαβε χώρα και συνδεόταν με επενδύσεις για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία. Ήταν πολύ επιτυχής η χρονιά, μετά μειώθηκαν τα αποτελέσματα και χρειάστηκε μεγάλη χρονική περίοδος και μεγάλη αναδόμηση για να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα. Άλλες πόλεις το πέτυχαν αμέσω. Η Λίλ, ε, ε, το πρόγραμμα Λίλ 3000, που απέρευσε από το ότι ήταν πολιτιστική ποτέ το 2008 ε, και είναι σημαντικό σημείο αναφοράς. Λοιπόν, στην έκθεση βλέπετε διάφορα παραδείγματα, αλλά τελικά αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ένας και μόνος τρόπος να πετύχει το σωστό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, ίσως δεν χρειάζονται όλες οι πόλεις αποτελέσματα τον τουρισμό, να το θέσω σαν βασικό στόχο. Λόγω μεγέθου και επενδύσεων κάποιε πόλει χρειάζονται τον κοινωνικό προγραμματισμό και το όφελο είναι η, διασύνδεση, η εκ νέου διασύνδεση διαφόρων κοινοτήτων. Κάποιε πόλει, λίγε πόλει μπορούν να πετύχουν ταυτόχρονα σε όλε τι πτυχέ. Τουρισμό, κοινωνικό τομέα, πολιτιστικό τομέα. Άλλε πόλει εστιάζονται περισσότερο σε έναν τομέα ή τα καταφέρουν καλύτερα σε έναν τομέα ή σε άλλο τομέα. Και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι αρνητικό. Θεωρώ ότι είναι σωστό να δεχτούμε ότι κάποιες πόλεις ήταν επιτυχέστατες όσον αφορά το τουριστικό μέτωπο, άλλες πόλεις δεν θεώρησαν ότι ήταν τόσο σημαντικό αυτό, ήταν πιο σημαντικό να υπάρχει κάποια διασύνδεση με τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς κλπ. Ναι. Για να αξιολογήσουμε την, ε, την, επιτυχία πρέπει να κρίνουμε αν πέτυχαν του αρχικού του στόχου. Αν στόχο ήταν να γίνει τουριστικό προορισμό μια πόλη και δεν το κατάφερε, πρέπει να καταλάβει η πόλη γιατί δεν τα κατάφερε. Thank you very much. I think it was... Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ συνοπτική παρουσίαση και πολύ χρήσιμη. Μας δώσατε πολλές χρήσιμες ιδέες για τα επόμενα χρόνια. Και θα υποφεληθούν και οι επόμενες υποψήφιες χώρες. Λοιπόν, είναι παρούσα η Κομισιόν. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο από εκείνους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλαμε να πούμε απλώς ότι ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο γιατί παρήγγειλε αυτή τη μελέτη και την δόκτορα Γκαρσία. Για μας ήταν επίσης χρήσιμη η μελέτη γιατί ε, έχει μακροχρόνια αντιμετώπιση. Από την Κομισιόν θέλω να επιμείνω στο τελευταίο που είπε η δόκτωρ Γκαρσία, δηλαδή ότι τελικά το σημαντικότερο για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι το πρόγραμμά της να συμπεριλαμβάνεται σε μια γενικότερη στρατηγική. Μίλησε για αστική ανάπτυξη. Δεν είναι πράγματι αυτό από τους κύριους στόχους όλων των πρωτευουσών. Είναι για τη Μασαλία, για την Κόσιτσε, αλλά για το Σαν Σεμπαστιάν όχι. Είναι ήδη βέβαια μια αρκετά γνωστή πολιτιστικά όλοι λόγω του φεστιβάλ κινηματογράφου. Ο στόχος της είναι μάλλον να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στις πολιτιστικές δραστηριότητες ή σε αυτήν την πολιτιστική δραστηριότητα που μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη σε αρκετά ελιτιστικό επίπεδο. Δεν έχουν όλες οι πόλεις λοιπόν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους, αλλά ευχαριστώ εκ νέου το Κοινοβούλιο που επέμεινε στις διαπραγματεύσεις να παραμείνει το κριτήριο αυτό στη νομική βάση. Γιατί αυτό που διαχωρίζει την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα με άλλες πρωτοβουλίες όπως την Αγγλική UK City of Culture που έχει περίπου παρόμοιους στόχους με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα η διαφορά είναι ότι βέβαια δεν έχει τόσο πολύ ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, λέει η πρόεδρος, αν στο Ηνωμένο Βασίλειο προσθεθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση και αν ποτέ υπάρξει ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως να ικανοποιηθούν και αυτά τα αιτήματα. Λοιπόν, υπάρχει εδώ σε αυτό το δημοσίευμα που σας δείχνω ολόκληρη η μελέτη. Ίσως έχει και περισσότερες πληροφορίες για την χωροταξία και την αστική ανάπτυξη και θα τη συζητήσει ελπίζουμε και το Συμβούλιο. Εμείς θέλησαμε να δώσουμε μάχη για τρεις στόχους την νοστική ε, ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή ταυτότητα κλπ. Ε, κερδίσαμε, όχι σε όλα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα την αφήσαμε τελικά. Η ευρωπαϊκή διάσταση άρκεσε. Ευχαριστούμε, περνάμε στο επόμενο σημείο. Απαλλαγή 12. Γενικός Προϋπολογισμός της Ένωσης. Ο Μόρτεν Λόκεγαρ θα μας κάνει την εισηγήσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όπως ξέρετε βέβαια ο ρόλος μας ως Κοινοβούλιο είναι κάθε χρόνο να χορηγούμε την απαλλαγή στην Κομισιόν για το προηγούμενο έτος μέσω μιας εξονυχιστικής εξέτασης του τρόπου δαπάνησης του προϋπολογισμού της από την Κομισιόν και η διαδικασία αυτή την αναλαμβάνουν γνωστοί και ικανοί συνάδελφοι οι οποίοι συμβουλεύονται όλες τις επιτροπές μεταξύ των οποίων και τη δική μας. Τώρα εξετάζουμε το 2012, φαντάζομαι ότι διαβάσατε όλη την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και την έκθεση πεπραγμένων της Κομισιόν και για τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Αν όχι τότε να σας κάνω μία σύντομη περίληψη. Στην έκθεσή μου δίνω συγκεκριμένε πληροφορίες για τα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, αθλητισμό, παιδεία και βλέπουμε πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα, αν κάτι είναι ασαφές ρωτάμε την Κομισιόν που οφείλεται η ασάφεια. Πρέπει να έχετε στο φάκελό σας την έκθεση και ιδιαίτερα έξι συγκεκριμένες παραγράφους χωριστές που σας ζητώ να τη σχολιάσετε αν θέλετε και κοιτάξτε ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν την ενωσιακή τεχνογνωσία αν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο δαπάνησε τα χρήματά της για αυτόν τον στόχο η Κομισιόν. Συνεργάστηκα και με τους Κιώδης βέβαια και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω κύριε Πρόεδρε. Αν έχετε σχόλια να τα ακούσω. fertig. Okay. So, äh, äh, Τον Ιανουάριο λοιπόν θα ψηφίσουμε. Όχι. Τροπολογίες μέχρι τις 15 ε, Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Ε, θέλει να μιλήσει η Κομισιόν επ' αυτού. Είναι κανείς εδώ. Έχει κάνει αντιρρήσει. Έχετε καμία αντίρρηση. Όχι. Όχι κανεί Α, καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επόμενο θέμα. 6. Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά. Πολιτιστικές και εκπαιδευτικέ πτυχές. Σαντιάγο Φίσας. Έκθεση πρωτοβουλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ντόρις. υπενθυμίζω καταρχάς τον ορισμό της λέξης γαστρονομία. Έχει διάφορες ε, έννοιες ε, σε σχέση με διάφορες πλευρές της διατροφής υγεία, ευχαρίστηση και ε, διαιτητική και κοινωνικές πλευρές, οικογενειακές πλευρές, πολιτιστικές, οικονομική σημασία απασχόληση και τουρισμός. Και φυσικά την αυστηρή γαστρονομική έννοια. Η απόλαυση ε, της βρώσης και πόσης. Η γαστρονομία ε, έχει όλες αυτές τις πλευρές. Παίζει λοιπόν μεγάλο ρόλο στην ποιότητα ζωής ε, των συμπολιτών μας. Αν, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Υπάρχει 1,2 δισεκατομμύριο, δισεκατομμύρια άτομα που είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Και περίπου το ίδιο, ο ίδιος αριθμός στοιχείων πάσχει από, ε, ατόμων πάσχει από, υπερσι, από υποσυντισμό. Και ε, από ό,τι μας λένε το 2040 περίπου ο μισός πληθυσμός θα έχει πρόβλημα ε, βάρους. Θα είναι δηλαδή παχύσαρκη. Επίσης στις ΗΠΑ προειδοποιούν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση παχυσαρκίας των παιδιών, θα υπάρξει μια γενιά που θα έχει προσδόκιμο ζωής ε, χαμηλότερο από την προηγούμενη γενιά. Δηλαδή, τα παιδιά θα ζουν λιγότερο από τους γονείς. Υπενθυμίζω ότι η παχυσαρκία είναι το πρώτο αίτιο θανάτου στον κόσμο. Και αυτό συνδέεται και με ένα όλο και πιο καθιστικό τρόπο ζωής, ε, ανενεργό αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά κινούνται λιγότερο, δεν πάνε με τα πόδια στο σχολείο, δεν παίζουν στο δρόμο, στα πάρκα. Κάθονται μπροστά στις βιντεοκονσόλες, στα βιντεοπαιχνίδια, το διαδίκτυο κλπ. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά αυτές τις γαστρονομικές αξίες και τη σημασία επίσης της σωματικής άσκησης. Έχουμε λοιπόν δύο προβλήματα, παχυσαρκία και καθιστική ζωή. Τι πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τις τάσεις αυτές που είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο. Το σχολείο πρέπει να παίξει ε, τον κυριότερο ρόλο, να αναλάβει τον πρώτο ρόλο σε σχέση με την οικογένεια που τον έχει τώρα σε πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτό το δίκτυο 10 χωρών ε, ιδρυμάτων για την ε, Διατροφή που προσπαθεί να ενημερώσει για τις καλές πρακτικές μεταξύ των χωρών αυτών και έγινε μια συνεδρίαση τον Απρίλιο 2010 στη Μαδρίτη για τη διατροφή στα σχολεία ε, σε όλη την Ευρώπη όπου μιλάμε για το πώς διδάσκεται η διαιτητική και το τι τρόφιμα παρέχονται στις σχολικές καντίνες. Και Αναφέρονται λοιπόν όλες αυτές οι εκπαιδευτικές πλευρές που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, αλλά και οι πολιτιστικές πλευρές και οι οικονομικές πλευρές της γαστρονομίας. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεσή μου. Στο τμήμα που ασχολείται με την εκπαίδευση καλούνται τα κράτη-μέλη να βάλουν στα προγράμματά τους, ε, τα σχολικά προγράμματα, ε, ε, μαθήματα για την γαστρονομική κουλτούρα, τις διαιτητικές συνήθειες, το μαγείρεμα και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και τα δίκαια του καταναλωτή στον τομέα αυτό. Οπότε πρέπει επίσης να υπάρχει και σωστή διατροφή, σωστά γεύματα στα σχολεία. Και στο κεφάλαιο αυτό μιλάμε επίσης για την αναγκαιότητα να υπάρχει επαρκής ε, αθλητισμός και σωματική άσκηση στα σχολεία. Επίσης η καλύτερη διατροφή βελτιώνει τη δυνατότητα ε, μάθησης των μαθητών και επηρεάζει τις διατροφικές του συνήθειες ε, μετέπειτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή επιμόρφωση και των καθηγητών για να μπορούν να διδάσκουν σωστά και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια για τα θέματα αυτά. Μετά μιλάμε στο πολιτιστικό τμήμα κυρίως για την ανάγκη να γίνει γνωστή η ποικιλότητα της ε, ευρωπαϊκής κουζίνας, να προωθήσουμε προϊόντα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς, να προωθήσουμε την τοπική γαστρονομική κουλτούρα και να μπει και στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Ήδη ορισμένα στοιχεία αναφέρονται. Λέμε στις πόλεις να υποβάλουν υποψηφιότητες για πόλη UNESCO της γαστρονομίας και επίσης αναφέρουμε ότι η γαστρονομία είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της εστίασης, της αγροδιατροφικής βιομηχανίας, του τουρισμού, της έρευνας και πολλά άλλα και κυρίως να προωθήσουν διατροφικές συνήθειες που να έχουν στόχο να διατηρήσουν την υγεία των καταναλωτών και να διατηρήσουν και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό η απόλαυση του φαγητού, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα. Ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων, βέβαια δεν είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, να δούμε μετά τι προθεσμίες έχουμε για να υποβάλουμε τροπολογίες για να το εγκρίνουμε το Φεβρουάριο νομίζω αλλά η γραμματεία θα μας πει πότε θα εγκριθεί η εκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σαντιάγο. Έχει ζητήσει ε, πρώτα απ' όλα η Έμα Μακλάκιν και μετά ο κύριος Τόκιος. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο σας πρώτα απ' όλα για το σχέδιο έκθεσης του. Συμπεριέλαβε πολλές από τις συστάσεις που εκφράσαμε και πολλές δικές μου και ευχαριστώ. μα αρέσει σαφέστατη δομή του κειμένου. Πολιτιστικές πτυχές, πτυχές εκπαίδευσης, εύληπτο το κείμενο και χαίρομαι επίσης και για τις πολιτιστικές πτυχές που αναφέρονται. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ αρμοδιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτιμώ πολύ το ότι εκτιμάτε την κοινωνική και πολιτιστική αξία της γαστρονομίας, το ίδιο πιστεύω, για τη γαστρονομική κληρονομιά, κυρίως να υποστηρίζουμε τις διάφορες ε, τοπικές εκδηλώσεις γαστρονομικού περιεχομένου. Οι τροπολογίες μου στο κομμάτι εκπαιδευτικό Πρέπει να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ αρμοδιοτήτων. Να σεβόμαστε την εκπαίδευση που θεωρείται αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρέπει να τονίσουμε την σημασία να μάθουν τα παιδιά για την γαστρονομική τους κληρονομιά όταν είναι πολύ μικρά. Αυτό θα τα βοηθήσει να καταλάβουν τη σημασία της διατροφής και των τροφίμων. Είναι ένα άλλο τμήμα του θέματος πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο επί των πολιτιστικών πτυχών και όχι τόσο επί της διατροφής, διότι δεν είναι τόσο αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Υπάρχουν άλλοι τομείς γαστρονομικοί που θα ήθελαν συμπεριληφθούν. Θα ήθελαν να συμπεριλάβουμε την προστιθέμενη αξία της γαστρονομίας όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την απασχολησιμότητα των νέων. Πολλοί νέοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας και ασχολούνται με τη γαστρονομία. Να τονίσουμε την αξία που έχει και είναι πολύ ισχυρό εξαγωγικό στοιχείο. Και έχουμε και θαυμαστούς ε, σεφ ε, στην ε, Ευρώπη. Είναι υπέροχη δουλειά που έκανε και ο Σφίσας με την έκθεση του και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί του στον τομέα αυτό και σε συνεργασία με τους κοιόδη συναδέλφους μου. Και εύχομαι υπέροχα Χριστούγεννα, πλούσια γαστρονομικά Χριστούγεννα. Uh, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζηλεύω τον κύριο Φίσας που ετοίμασε με τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση. Είμαστε υπερήφανοι για τη γαστρονομία μας στην Τρανσιλβανία, στην Ουγγαρία. Η γαστρονομία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας κάθε χώρας, κάθε λαού. Και όπως και η εινολογία εξάλλου. Έχουμε πάρα, πολύ καλά κρασιά στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Όταν είχαμε πάει επί τόπου, πάντα είχαμε εκτιμήσει τα εστιατόρια, τα κρασιά. Είναι αναφυσβήτητο λοιπόν ότι η γαστρονομία αποτελεί τμήμα των μέσων που διαθέτουμε για να γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας. Η γαστρονομική κληρονομιά των λαών παίζει σημαντικό ρόλο. Σήμερα λοιπόν όταν η αμερικανική κουλτούρα κατακλίζει την Ευρώπη με προϊόντα fast food είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτή την γαστρονομική κουλτούρα μας. Είμαστε Ευρωπαίοι και θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη την κληρονομιά κάθε χώρα σε κάθε λαού. Κάτι που αναφέρατε. Αυτό λοιπόν το μέσο, ε, αυτά τα μέσα που αναφέρονται μπορεί να διευκολύνουν την όλη διαδικασία και το πρόγραμμα αυτό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μπορεί να συμβάλλει στην όλη διαδικασία. Τα θέματα είναι αλληλένδετα λοιπόν. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει μια κοινωνική πτυχή που σχετίζεται κατά πολύ με τη γαστρονομία. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε φτώχεια, ε, Έχουμε τους Ρωμά. Υπάρχει μια κοινωνική πτυχή πάρα πολύ σημαντική στο θέμα που συζητούμε. Είναι πολύ μακριά αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια και στην απομόνωση από το γαστρονομικό κόσμο των σεφ που συζητούμε. Υπάρχουν εκατομμύρια που ζουν σε, άκρα ένδια. Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη, να σκεφτούμε τι δυνατότητες έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Δεύτερο, η παράδοση και η υγεία. Η παραδοσιακή κουζίνα δεν είναι πάντα και πιο υγιής. Σε εμά, στην Ουγγαρία, οι παλιοί είχαν μια διαφορετική γαστρονομική κουλτούρα που δεν ήταν τόσο υγιής. Πρέπει να αναπτύξουμε τις παραδόσεις, τις γαστρονομικές και να τις κατευθύνουμε προς την υγεία, να υπάρχει συνδυασμός παράδοσης με σωστή διατροφή. Να είναι πιο υγιής έτσι η κουζίνα μας και πιο ισορροπημένη. Εύχομαι καλό κουράγιο και καλή τύχη στο κύριο Σαντιάγο Φίσας και περιμένουμε την οριστική εκδοχή της έκθεσής του. Τελική μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Τούρκους. Η κυρία Σάντσες Σμιθ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Σαντιάγκο Φίσα για την έκθεσή του με σημαντικό νομίζω θέμα γιατί η γαστρονομία βρίσκεται στο κέντρο των ενδιαφερόντων πολλών και καμιά φορά μπορούμε να πούμε ότι παραγνωρίστηκε στον 20ο αιώνα ενώ είναι σημαντική πτυχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έχει και τουριστική πτυχή και έχει και υγειονομικό ενδιαφέρον. Ε, ακούστηκαν οι αριθμοί. Μόνο σας δώσω κι άλλο. 35 εκατομμύρια άνθρωποι το 2005 πέθαναν από μη μεταδοτικές ασθένειες αλλά συνδεόμενες με έλλειψη γυμναστική, γύμνασης ή οφειλόμενες στη διατροφή, σε κακή διατροφή. Η σημασία λοιπόν της σωστής διατροφής είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να αρχίζει η επιμόρφωση από αυτού από την νεαρή ηλικία, παιδική ηλικία και η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει πολλά στα σχολικά προγράμματα ας πούμε για την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, το School Food Scheme ας πούμε, που εφαρμόστηκε στη Γαλλία με άλλο γαλλικό τίτλο διότι έχουμε αρκετά διαφοροποιημένη γεωργία στην Ευρώπη και μπορούμε να αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Επίσης σημειώνω την πλευρά της ειδονής που σημείωσε ο κύριος Φίσας για την ε, γαστρονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να υποστηρίξει όλα τα σχετικά προγράμματα και την θεία ιδίω για την συνέχιση της γαστρονομικής κληρονομιάς, την πρόθεσή της, τη μετάδοση των γνώσεων και την υποστήριξη πρωτοβουλειών. Πολύ θα γνωρίζετε την οργάνωση slow food που αντιτίθεται στο fast food. Ιδιαίτερα για τα σχολεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως το Zardene Call. για να καταλαβαίνουν τα παιδιά καλύτερα από πού προέρχονται τα τρόφιμα και να γνωρίζουν και τα ωφέλιμα τρόφιμα. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλα θετικά στοιχεία της γαστρονομίας που δεν θα τα αναφέρω όλα, το, τουριστική πτυχή, η γαστρονομία είναι τμήμα των δημιουργικών αυτών τομέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μήπως κανείς από την Κομισιόν θέλει να σχολιάσει, όχι. Ο Σαντιάγος. Ευχαριστώ, Ντόρις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση. Φυσικά θα είναι ευχαρίστη συνεργαστώ με την Έμα Μακλάρκιν, όπως και στην έκθεση που είχαμε για... και για άλλα θέματα. Πρέπει οπωσδήποτε να αποτιμήσουμε όλες τις πλευρές της γαστρονομίας τη σχέση με τη φιλοξενία, τον τουρισμό, τους νέους, πολύ καλή ιδέα. Να τονίσουμε την ιδέα των μεγάλων σεφ που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Χωρίς να υποτιμούμε την γαστρονομία σε άλλες υπήρους, είναι ένα από τα μεγάλα προσόντα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Τώρα για τη διατροφή στα σχολεία κάνουμε απλώς συστάσεις. Γνωρίζω σαφώς ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική αρμοδιότητα. Στη χώρα μου συγκεκριμένα είναι αρμοδιότητα των ε, αυτονόμων κοινοτήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον να μάθουν τα παιδιά αυτές τις βασικές γνώσεις για θέματα διατροφής. Έγινε ένα μεγάλο σεμινάριο για το θέμα αυτό στη Μαδρίτη ε, και εκεί η προσωπικότητα του κυρίου Φουστέρ που εργάζεται στη Νέα Υόρκη είπε ότι έκανε μια σειρά από δοκιμές με παιδιά από την Κολομβία και η γνώση για το πώς πρέπει να τρώει κανείς σωστά πρέπει να μεταδοθεί σε πολύ νέα ηλικία ακόμη και παιδιά τριών-τεσσάρων ετών τότε είναι που είναι εύκολο να τους ε, να μάθουν λοιπόν πώς να τρώνε σωστά, να έχουν τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον τους. Και η παρέμβαση του φίλου Τόκες ε, τόνισε αυτό που συζητήσαμε, η γαστρονομία και πολιτισμός και βοηθάει επίσης οπωσδήποτε και την ένταξη μιας σειράς εθνικών μειονοτήτων. Μπορεί να βοηθήσει και εδώ. Και στην Μαρή Τερέζ βεβαίως βάλαμε το θέμα του αργού φαγητού, slow food στην έκθεση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που αναφερόμαστε σε αυτό. Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε αυτή την αντίθεση με το fast food με χαρά λοιπόν θα συνεργαστώ με τους σκιώδεις και επίσης να εξετάσω τις τροπολογίες που θα μπορούσαν να υποβληθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Λοιπόν, 16 Ιανουαρίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών και θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο 7 ας περάσουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Θεάτρων. ETC, European Theatre Convention, η οργάνωση αυτή δημιουργήθηκε το 1988, είναι πανευρωπαϊκό δίκτυο που αντιπροσωπεύει τον ε, τομέα των ε, δημοσίως επιδοτουμένων θέατρων σε 25 χώρες θέλουν να προωθήσουν το σύγχρονο θέατρο, ανταλλαγές ε, και κινητικότητα καλλιτεχνών στην Ευρώπη και ευρύτερα και επίσης θέλει να εκτελέσει προγράμματα κατάρτισης και άλλες δυνατότητες κατάρτισης στα πλαίσια της διαβίου μάθησης και να βοηθήσει τους νέους δημιουργούς στον τομέα του θεάτρου. Στο παρελθόν το ETC ε έχει λάβει επιδότηση και από το δικό μας προϋπολογισμό. Καλέσαμε τον κύριο Γκέργκορ και τον κύριο Ραγκόνη. Έχουν ο καθένας από 10 λεπτά το λόγο. Παρακαλώ περάστε μπροστά.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 it works. Okay? So. It works? Yeah. Okay. Yeah, you should, you, sh you should speak. Dubravka Vergoc, it seems that she... Dubravka Vergoc. Είστε από την Κροατία. Ναι, είμαι από την Κροατία. Ευχαριστώ κυρία Πακ που μας καλέσατε να μιλήσουμε για το θέατρο. Μετά την γαστρονομία πολύ καλό να μιλήσουμε για το θέατρο. Αν και βέβαια πρώτα πάει κανείς στο θέατρο και μετά τρώει. Χαίρομαι που μπορούμε να μιλήσουμε για το θέατρο, για το θέατρο γιατί περνάει δύσκολη περίοδο λόγω της ύφεση στις χώρες μας. Άρα έλλειψη πιστώσεων για την τέχνη άρα και για το θέατρο. Αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το θέατρο στη ζωή μας, όπως ήταν για τόσους αιώνες. Πρέπει να πολεμήσουμε για να έχει τη θέση που του αρμόζει. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Πολιτισμού είναι νομίζω οι κατάλληλοι φορείς να παλέψουν για το θέατρο. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η Σύμβαση για το Θέατρο, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Είμαστε λοιπόν οι παλιότεροι, το παλιότερο και ευρύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Δημιουργήθηκε το 1988, τότε συμμετείχαν τρεις χώρες, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία. 25 χρόνια αργότερα, σήμερα δηλαδή, έχουμε πάνω από 40 θέατρα μέλη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, από τη Φιλανδία στην Κύπρο, και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πάνω από 20 χώρες ε, συμμετέχουν και εκφραζόμαστε σε 22 γλώσσες. Εργαζόμενοι στα θέατρά μας, στα θέατρά 11.000 εργαζόμενοι. Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε 16.000 παραστάσεις με 8 εκατομμύρια θέατες. Η οργάνωσή μας βασίζεται για να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία, την κινητικότητα και τον ε, διαπολιτιστικό διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεάτρων και χωρών. Είναι επίσης μια πλατφόρμα για επαγγελματικές ανταλλαγές αυτών που συμμετέχουν στον τομέα για να δημιουργηθεί σύγχρονο θέατρο και γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και να προωθήσει και να εκπροσωπήσει τον τομέα του δημοσίου θεάτρου στην Ευρώπη. Προτεραιότητα στην εργασία μας είναι αυτή η συνεργασία, είναι τα διαπολιτιστικά προγράμματα συνεργασίας. Τι θέλουμε, να βοηθήσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στο θέατρο, να συμμεριστούμε τις βέλτιστες πρακτικές μέσω συνδιασκέψεων, συναντήσεων, επαγγελματικών ανταλλαγών λοιπόν, Επίσης μια νέα κοινή στρατηγική για ανάπτυξη του κοινού. Να προωθήσουμε την πολυγλωσία, γιατί το θέατρο, ξέρετε, βασίζεται στην προφορική έκφραση. Παρουσιάζουμε έργα σε 22 γλώσσες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν ανταλλαγές από αυτών των θεμάτων. Κάνουμε πολλά για την επιμόρφωση στον τομέα του θεάτρου Έχουμε προγράμματα συνεργασίας μεταξύ της οργάνωσής μας και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν σχέση με το θέατρο. Ποιο είναι το κύριο πρόγραμμά μας που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρόγραμμα 2004-2013, ε, ε, είναι η τέχνη της γύρανσης. Συνεργάζονται οκτώ θέατρα και από τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Θέλουμε περισσότερη συνεργασία διαπολιτιστική που να βασίζεται σε θέατρο, στο θέατρο και σε μορφές ντοκιμαντέρ. Μας βοηθάει η Ετέλα Τνάν που είναι θεατρική συγγραφέα 87 ετών. Θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε διάφορες πλευρές της τέχνης της γύρας, οικονομικές, κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές, πολιτικές. Γιατί διαπιστώνουμε ότι το κοινό μας ε, κατά μέσο όρο είναι άνω των 60 και το θέατρο δεν έχει λάβει τόσο πολύ υπόψη το γεγονός ότι οι θεατές μας είναι ε, ηλικιωμένοι και ότι οι ηλικιωμένοι υπάρχουν και κάναμε κάτι διαφορετικό τα τελευταία χρόνια ήταν το πρόγραμμα για την Ευρώπη των νέων Είχαμε δύο τέτοια προγράμματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι ε, μια πρωτοβουλία που λέγεται η ε, Νέα Ευρώπη, ε, πολυγλωσσική δημιουργία και εκπαίδευση. Ανεβάζουμε λοιπόν πολύγλωσσα έργα σε συνεργασία με νέους επαγγελματίες του κλάδου. Στόχος να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων στο θέατρο και τον πολιτισμό και να υπάρχει ένας χώρος οι νέοι μας να ε, αμφισβητήσουν τις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλαμε να συνδέσουμε το σχολείο με το θέατρο, την εκπαίδευση με τον πολιτισμό. Οι περισσότερες παραστάσεις έγιναν στα θέατρα, στα σχολεία, με συγχωρείτε, είτε με κοινό μαθητών στα θέατρα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι συνεργασία 8 ε, θεάτρων. Οργανώσαμε 16 παραστάσεις. Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας σε δύο φεστιβάλ στο Στρασβούργο και το Βερολίνο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και είχαμε επίσης μια κατασκήνωση στο Βερολίνο στα πλαίσια αυτά. Συμμετείχαν 400 επαγγελματίε, 17 δημόσια θέατρα, 12 χώρες και 40.000 νέοι Ευρωπαίοι ε, συμμετείχαν ως κοινό και δημοσίευσαμε και ένα βιβλίο με τα θεατρικά έργα. Εδώ βλέπετε κάποια εικόνα από τις παραστάσεις. Μετά είχαμε το πρόγραμμα «Η Νέα Ευρώπη 2», ίδιος τίτλος, αλλά παρουσιάσαμε τέσσερα έργα μεταφρασμένα σε οχτώ γλώσσες οι πρεμιέρες έγιναν σε ευρωπαϊκά θέατρα. Οργανώσαμε και ένα φεστιβάλ τον περασμένο Μάιο στο Βερολίνο υπό την αιγίδα της κυρίας Πάκα και της Επιτροπής σας. Επίσης, κάναμε και την κατασκήνωση των νέων ταλέντων της Ευρώπης για να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές ιδεών και να συνδέσουμε τους νέους με το θέατρο. Επίσης, έχουμε και το πρόγραμμα το Διεθνές Φόρουμ Νέων για το Θέατρο, που κάθε χρόνο γίνεται στο Bad Hersfelder στη Γερμανία. Συναντιόνται οι νέοι από διαφορετικές χώρες και για πρώτη φορά εργάζονται μαζί για το θέατρο, για να γνωριστούν, να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους στην Ευρώπη σήμερα. Το πρόγραμμα αυτό οργανώθηκε και το 2012 και πήρε ένα βραβείο στη Γερμανία για την καλύτερη ε, προβολή ιδεών, ένα βραβείο της γερμανικής κυβέρνησης. Τι άλλο κάνουμε. Πολλές ανταλλαγές ε, του προσωπικού των θεάτρων, τεχνική για παράδειγμα από τον Γκέλζεν Κίρχεν έρχονται στο Ζάγκρεπ, δουλεύουν ένα μήνα. Έχουμε επίσης ε, άλλου από τι δημόσιε σχέσεις των θεάτρων και άλλου. Έχουμε και ένα φεστιβάλ για νέους ε, καλλιτέχνε, γιατί θεωρούμε ότι στην Ευρώπη δεν θα έχουμε πρόβλημα με το κοινό, αλλά δεν θα έχουμε και καλλιτέχνες ε, λόγω κρίση. Δεν έχουν δυνατότητα να εργαστούν οι νέοι στο θέατρο και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Έχουμε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ για νέους σκηνοθέτες. Ήταν ε, ε, ευρείας διάστασης ε, φεστιβάλ στην Biennale του Βισμπάντεν. Επίσης έχουμε διάφορες ανταλλαγές μεταξύ δραματικών σχολών. Ανταλλαγών μεταξύ δραματικών σχολών και των θεάτρων μελών μας. Από το 2012 αυτό που κάνουμε και θεωρούμε σημαντικό είναι για το Ευρωπαϊκό Θέατρο είναι να αυξηθεί το κοινό μας. Κάνουμε διάφορες ε, μελέτες σε 10 χώρες, μεταξύ των μελών μας αυτές τις χώρες. Σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα θέατρα, είχαμε 1.745.000 θεατές. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, γιατί μόνο 10,2% από αυτούς τους περίπου 2 εκατομμύρια ατόμων δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε παραστάσεις, θα πάνε δηλαδή να δουν παραστάσεις ε, στο εξωτερικό αλλά ακόμη και μεταξύ του κοινού μιας πόλης μόνο 3,3% είπαν ότι θα πάνε να παρακολουθήσουν παραστάσεις άλλων θεάτρων. Κάποιοι βέβαια έρχονται για τα φεστιβάλ αλλά όχι τακτικά και παρά το ότι υπάρχουν υπότιτλοι όλο και περισσότεροι δεν είναι ακόμη επαρκές, ποσοστό, ε, επαρκές το ποσοστό υποτιτλισμού άρα δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσουν ε, κάποιοι παραστάσεις σε άλλη γλώσσα. Αλλά αυτό που είναι πολύ πιο ενθαρρυντικό είναι κάτι που μας εξέπληξε ακόμη και μας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή περισσότεροι ε, παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις παρά ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έχουμε παραδείγματα εδώ από τη Γερμανία και την Κροατία. Στη Γερμανία το θέατρο που λαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις είχε 19 εκατομμύρια θεατές, ενώ μόνο 13 εκατομμύρια πήγαν σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια της Bundesliga. Καλό για το ποδόσφαιρο, συγγνώμη, καλό για το θέατρο, όχι τόσο καλό για το ποδόσφαιρο. Στην Κροατία είχαμε 1,5 εκατομμύρια θεατές στο θέατρο το χρόνο, ενώ μόνο 30.000 πηγαίνουν ε, στα μάτς. Ενώ όπως ξέρετε η Κροατία είναι πολύ πιο γνωστή ε, για το ποδόσφαιρό της και όχι για το θέατρο της. Άρα είναι θαρρυντικό αυτό. Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Θέλουμε να εστιάσουμε σε τρία θέματα. Πρώτον, η ενεργός γύρανση Θέλουμε να συμμετάσχουν οι ηλικιωμένοι, να έρχονται στο θέατρο, να συμμετέχουν και θέλουμε να κάνουμε και έρευνα για τη θέση του ηλικιωμένου στην κοινωνία μας. Στα πλαίσια και της αύξησης του κοινού μας φυσικά. Αλλά και για να υπάρχει διαβίου μάθηση για τους ηλικιωμένου. Δεύτερον, το εργαστήρι για το Ευρωπαϊκό Θέατρο πρέπει να ψάξουμε για νέες θεατρικές μορφές να επανακαθορίσουμε τη θέση των θεάτρων ως θεσμών στην εποχή μας. Το εργαστήρι λοιπόν θα είναι πλατφόρμα έρευνας στις πόλεις, στις κοινωνίες μας για ανάπτυξη νέων μορφών στο δημόσιο χώρο, να έρθουμε σε επαφή με νέο κοινό. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια μελέτη μεταξύ των μελών μας για αύξηση του κοινού Έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία για το κοινό μας στην Ευρώπη και τα μέλη μας θέλουν να αναπτύξουν στρατηγικές marketing, να προσεγγίσουν το κοινό, γιατί αν επιτύχουμε στην Ευρώπη αυτό που γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, στη Νέα και για παράδειγμα τα τελευταία 10 χρόνια το κοινό είναι μόνο άνω των 60. Δηλαδή σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας θεατής. Εμείς ως δίκτυο πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά και σε βάθος αυτό το πρόβλημα. Η προσπάθεια λοιπόν να αυξήσουμε το κοινό είναι να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας. Γιατί είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με εσά, γιατί θέλουμε να υπάρξει επαφή μαζί σας, θέλουμε να υπάρχει διάλογος, εταιρική σχέση μεταξύ του δικτύου μας και των ευρωβουλευτών να επανακαθορίσουμε το ρόλο μας ως δημοσίου θεάτρου, δημοσίου θεσμού, ούτως ώστε να αλλάξουμε τα πρότυπα κατανάλωση πολιτισμού και ποια θα μπορούσε να είναι η διάδραση μεταξύ του θεάτρου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς πρέπει να παλέψουμε για το θέατρο την εποχή μας. Να μην συνεχιστούν οι τάσεις που διαπιστώνουμε τώρα, μείωση των επιδοτήσεων σε τοπικό επίπεδο, διότι έτσι ε, το θέατρο δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό που κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι πολύ καλά ότι στο Βερολίνο όταν προείδευα εκεί ήταν η ώρα της συζητήσεων και παρακολούθησα κάποιες παραστάσεις των νέων ήταν υπέροχα. Πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά. Δεν είσαστε ακόμα παντού. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν συμμετέχουν. Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ζεγοβίνη και λοιπά υποψήφιες χώρες και Αλβανία λένε ότι ενδιαφέρονται. Άρα αυτή είναι μια γέφυρα για αυτές τις χώρες να είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να βρείτε τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις δραστηριότητες σας περαιτέρω και υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη που σας παρέχει πολλές δυνατότητες για διάφορα προγράμματα. Ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε αργότερα. Με ποιο τρόπο χρηματοδοτήστε. Διότι δεν θα πάρετε όλα τα χρήματα από εμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα μπορείτε να δώσετε την απάντηση. Τώρα η Χέλγα έχει κάτι να πει. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπατε, ότι θέλετε να προωθήσετε την ευρωπαϊκή συνεργασία. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα πράγματα για τα σχέδιά σας. Τι πιστεύετε θα κάνετε τα επόμενα χρόνια σχετικά με αυτό. Ήδη αναφερθήκατε στο πρόβλημα των επιδοτήσεων που στο εθνικό επίπεδο μειώνονται συνεχώς. Άρα, ποιο είναι ο στόχος σας. Τι θα θέλατε να δείτε να συμβαίνει τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταβάρες έχει το λόγο. Είναι εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούνε οι διερμηνείς δυστυχώς. Συγγνώμη. Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ και είπε και η κυρία Πακ, δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στο ETC. Ε Τι σχέδια έχετε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με τα εθνικά θέατα των κρατών μελών και με κάποια άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Έμα. Χαίρομαι που άκουσα αυτά που είπατε. Εξέτασα την ιστοσελίδα σας. Με το Nottingham Playhouse συνεργάζεστε στην εκλογική μου περιφέρεια. Χαίρομαι που συνεργάζεστε μαζί τους και προωθείτε τα όσα γίνονται στην Ευρώπη. Θέλω να καταλάβω πώς ξέρετε τους ακροατές τον αριθμό των θεατών μάλλον βασίστε στα εισιτήρια που κόβονται. Αν πάει κανείς στο θέατρο πάει συνέχεια. Και ανησυχώ για εκείνους που δεν εκτίθενται στο θέατρο καθόλου. Πώς μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε αυτούς που δεν πήγαν στο θέατρο να πάνε στο θέατρο. Να απαντήσω και μετά θα δώσω το λόγο στο ΣΕΣΠΟΝ αντιπρόεδρο ΕΕ, για τη χρηματοδότηση. Από τα μέλη μας χρηματοδοτούμεθα συν χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό 2007-2013 για τη δικτύωση και για προγράμματα και στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασία και σχέδια και προγράμματα. Να πω κάτι. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε στη χώρα σας που υπάρχουν θέατρα, ε, να έρθετε σε επαφή με τα θέατρα και να πείτε να γίνουν μέλη μας και να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Διότι αν μεγαλώσουμε σημαίνει ότι μπορούμε όλοι μαζί να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε εποχή ύφεσης και οικονομικών προβλημάτων τώρα είναι πιο σημαντική συνεργασία στο θεατρικό τομέα. Ο ΣΕΣ... Και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω ως αντιπρόεδρος της συνέλευσης αυτής Πριν από μερικές μέρες μάθαμε τις σχετικές προτάσεις σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι το θέατρο ακόμα και από οικονομικής απόψεως θεωρείται αρχαϊκή δραστηριότητα διότι ο αριθμός των εργαζομένων εκεί δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνολογία. Αυτό βέβαια είναι και ένα θετικό στοιχείο για την Ευρώπη γιατί είναι τέχνη που προϋποθέτει ανθρώπινη επαφή και επαφή μεταξύ κοινού και επαγγελματιών. Ως οργάνωση θα ήθελα να σας αναφέρω και μερικά από τα προβλήματά μας, από τις ανησυχίες μας, που ίσως να μπορούσατε κι εσείς να τις συζητήσετε. Πρώτον, για την κυκλοφορία των θεαμάτων και το φόρο τη προστιθέμενης αξίας τους. Ξέρω ότι δεν είναι αρμόδια η δική σας επιτροπή, αλλά είναι από τα σημαντικότερα μας προβλήματα με τα υπόλοιπα χρηματικά προβλήματα που έχουμε στις διάφορες χώρες και μάλλον κάποια βελτίωση σε αυτό το θέμα θα βελτίωνε την ε, κυκλοφορία των θεαμάτων. Η κινητικότητα εξάλλου είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αντικείμενο προγραμματισμού ή κάποιας πολιτικής ή οικονομικής στήριξης από την Ευρώπη. Τρίτον, οι μηχανισμοί πρόσβασης στα θεάματα υποτιτλισμός, ταυτόχρονη μετάφραση, όλα αυτά δεν στηρίζονται από τα ευρωπαϊκά κράτη ούτε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, η επαγγελματική εμπειρία και επαφές, δίκτυα κινητικότητα των θειάσεων, όλα αυτά τέθηκαν ιδίως μετά την ένταξη των ε, χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και κατέληξαν σε αύξηση του κοινού και των θεατών και αυτά όλα είναι ίσως ορισμένες ιδέες που εμάς μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και που Ίσως να μπορούσαμε να συνεργαστούμε από αυτόν και με την Ευρώπη. Νομίζω. Η προσέγγιση σας που μας περιγράψατε αφορά και την διαβίου μάθηση για νέους και την δική τους κινητικότητα κατά πόσον ενδιαφέρονται για το θέατρο. Εάν οι θεατές είναι όλοι της ηλικία μου Αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε κάποτε να μάθουμε τι είναι το θέατρο, να το συνηθίσουμε. Οι νέοι ήδη λοιπόν στο σχολείο πρέπει να φροντίσουμε να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για το θέατρο. Όποιος κάθεται μόνο μπροστά στον υπολογιστή του βέβαια δεν θα πάει στο θέατρο. Θα πρέπει λοιπόν στον τομέα της εκπαίδευσης ε, να στραφείτε. Οπωσδήποτε λοιπόν να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα Erasmus ΣΥΝ, που είναι η συνέχεια του διαβίου μάθησης, το τμήμα του που αφορά τους νέους. Άρα να έρθετε σε επαφή με την Κομισιόν για να δείτε πώς θα πρέπει να διατυπώσετε, να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα για να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι και το πρόγραμμα αυτό αλλά και άλλα προγράμματα όπως η Δημιουργική Ευρώπη θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα μόνο βέβαια. Στη Δημιουργική Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που αφορά τα μέσα και τον κινηματογράφο. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Αλλά δεν περιέχεται τίποτα για το θέατρο ή σχεδόν τίποτα. Το θέατρο στον τομέα αυτού του προγράμματος δεν παίζει κανένα ρόλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επιχειρήσουμε στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης να υποστηρίξουμε και τέτοια προγράμματα μαζί με το Έρασμος ΣΥΝ. Στα πλαίσια του Έρασμος ΣΥΝ. Να το σκεφτείτε λοιπόν και είμαι βεβαία ότι η Κομισιόν έχει επαρκείς υπαλλήλου που μπορούν να σας βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Αλλά όπως σωστά είπατε ή όπως σωστά είπε η συνάδελφος Έμα και στις δικές μας εκλογικές περιφέρειες εμείς πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για το θέατρο. Αλλά όλα τα θέατρα έχουν το ίδιο πρόβλημα, δεν έχουν χρήματα. Ίσως λοιπόν μέσω της συνεργασίας να υπάρξει περισσότερη διατομιακή προσέγγιση και διαπολιτιστική προσέγγιση που να βοηθήσει ε, τους ε, θεατές ε, να παρακολουθήσουν παραστάσεις σε άλλη γλώσσα. Στην όπερα γίνεται πολύ γιατί τα περισσότερα, οι περισσότερες όπερες είναι στα Ιταλικά και τις παρακολουθούμε. Μέσω υποτιτλισμού, μέσω συγχρονισμού είναι πολύ ακριβό και δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει για τον κινηματογράφο που πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια πολυγλωσσίας. Είναι δυνατό λοιπόν και για τα δύο προγράμματα να υποβάλλετε αιτήσει για χρηματοδότηση, αλλά παρακαλώ προηγουμένως να ενημερωθείτε για το πώς πρέπει να τις διατυπώσετε. Άλλος τις; Α, η Κομισιόν. Α, όχι. Α, όχι η Κομισιόν. Α, κανείς. Μάλιστα. Άλλος τις... Θέλετε πάλι το λόγο εσείς. Ντομπράβκα. Ήθελα απλώ να σας ευχαριστήσω για αυτό που είπατε γιατί τον αγώνα με την, για τη δημιουργία της δημιουργικής Ευρώπης θα τον χάσουμε, κινδυνεύουμε και πρέπει ο αγώνας να γίνει πιο έντονος από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Εάν τώρα δεν έχουμε καμία θέση στο νέο πρόγραμμα της Κομισιόν, φανταστείτε τι θα γίνει μετά από 7 χρόνια. Αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να αγωνιστούμε για να βρούμε έναν τρόπο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλα τα προβλήματα που έχουμε και αναφέρθηκαν σήμερα. Είναι το θέμα της νεολαίας, δηλαδή δεν έχουν οι νέοι ηθοποιοί θέση αυτή τη στιγμή δημιουργική γιατί δεν υπάρχουν χρήματα η τέχνη αυτή τη στιγμή γίνεται, μπαίνει στο περιθώριο. Εμείς πού θα μπούμε, τι θα γίνουμε. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από πριν λοιπόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη δική σας βοήθεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το κοινό, οι νέοι, το θέατρο είναι σημαντικά πράγματα και πρέπει να κρατήσουμε το θέατρο ζωντανό και για το μέλλον. Είναι εδώ η κρίσιμότερη στιγμή νομίζω. Έχω μία αντίρρηση. Το νόιο πρόγραμμα δεν ενδιαφέρεται λιγότερο για τη δουλειά σας από ότι το προηγούμενο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Από ό,τι θυμάμαι, ε, επιμείναμε να μπει η λέξη θέατρο και η λέξη καλλιτέχνες που δεν αναφέρονταν ήδη. Φυσικά ε, η Δημιουργική Ευρώπη ε, είναι συνδυασμός δύο προγραμμάτων, το πρόγραμμα πολιτισμός και το πρόγραμμα για τα μέσα. Δεν θα πρέπει να νομίζετε ότι έχετε τώρα λιγότερες δυνατότητες από ό,τι πριν. Έχετε τουλάχιστον τις ίδιες, ίσως λίγο περισσότερες. Γιατί εκπεφρασμένα αναφέραμε αυτά που προανέφερα. Βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα που υπέβαλε η Κομισιόν, αλλά το ε, εκτελεί ε, και το ενέκρινε το Συμβούλιο και εμείς. Εμείς ε, λάβαμε την πρόταση που μας υπέβαλε η Κομισιόν, την τροποποιήσαμε εν μέρη και είμαστε συνυπεύθυνοι. Αναφέρεται το θέατρο. Και εφόσον αναφέρεται μπορεί να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα για το θέατρο. Εάν κάνετε φεστιβάλ για παράδειγμα στα πλαίσια του προγράμματος θα μπορούσατε να κάνετε αίτηση χρηματοδότησης. Υποστηρίζουμε και φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν φυσικά θα χρηματοδοτηθείτε κάθε φορά, γιατί βεβαίως υποβάλλονται πολλές, ε, πολύ περισσότερες αιτήσει από ότι έχουμε πιστώσεις. Αλλά θα πρέπει όλοι στα πλαίσια των ήδη δημιουργηθισών ε, ε, δυνατοτήτων να επιχειρήσετε μέσω της Δημιουργικής Ευρώπης και μέσω του Erasmus Plus να, συν να χρηματοδοτηθείτε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη ζήτηση και εύχομαι να ε, υποστηριχθείτε την επόμενη 7 ετία και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε κάπου είτε στη, στο Ζάγκρεπ είτε στο Πάκαουα οπουδήποτε. Επόμενο θέμα της συνεδρίασής μας είναι είναι συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ λοιπόν όλους όσους δεν ε, ε, δικαιούνται να συμμετάσχουν στις συνεδρίες των συντονιστών να εξέλθουν.